Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώ ήρθατε σε αυτήν την τελευταία μα συνεδρίαση πριν από τι Χριστουγεννιάτικε διακοπέ. Πριν δώσω το λόγο στον Επίτροπο, στο σημείο 1 που μιλάει για την έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Να σας πω ότι η κυρία Σημέρα θέλει το δικό της το σημείο για τις ίσες ευκαιρίες και τα δικαιώματα της γυναίκας να το εξετάσουμε πριν από το σημείο 5. Αν δεν έχετε αντίρρηση λοιπόν, αυτό θα κάνουμε. Η κυρία Μωράρη Σαπιέ είπε ότι το δικό της το σημείο για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων εξεταστεί πριν από τις 4 και 5. Θα προσαρμόσουμε συνεπώς, εάν χρειαστεί, ανάλογα την ημερήσια διάταξη. Το σημείο 2, ανακοινώσει της Πρόεδρου, Α το αφήσουμε για μετά την ε, συνάντησή μας εδώ με τον Επίτροπο για να μην το καθυστερήσουμε άλλο. Οπότε θα δώσω το λόγο αυτής αμέσως στον Επίτροπο. Αλλά να σας εξηγήσω λιγάκι για ποιο λόγο εμείς εδώ στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων θελήσαμε να έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο και μετά θα, θα δώσω το λόγο στη συνάδελφο Γιούτα Στάινρουκ που είναι η συγγήτρια για το πρόγραμμα για την κοινωνική ελεγχή και την καινοτομία που υποβάλλει προφορική ερώτηση στην Επιτροπή. Κύριε Επίτροπε, θα θυμόσαστε ότι πολλές φορές μέχρι τώρα έχουμε επιστήσει την προσοχή σας στην διάρθρωση που υπάρχει ανάμεσα στην μεταρρύθμιση του Γιούρες που προβλέπετε εσείς και την συνθήκη της Λισαβόνας που τροποποιεί τη νομική βάση βάσει της οποίας ε, καθορίζεται το Γιούρες και δίνει περισσότερες αρμοδιότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι δύο επιστολές που σας στείλαμε έμειναν αναπάντητες. Ανησυχούμε λοιπόν για τη συνέχεια της διαδικασίας και μάλιστα από νομική άποψης, αυστηρά νομική, που έχει να κάνει με τη θέση σε ισχύ της συνθήκη της Λισαβόνας, σχετικά με το ενδεχόμενο μεταρρύθμισης του Γιούρε χωρίς συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και το άλλο είναι η διάρθρωση που σας είπα την, ε, ανάμεσα στη μεταρρύθμιση που προβλέπετε και τις εξελίξεις στη συναπόφαση για το πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία. Θα δώσω το λόγο όμως στην εισηγήτριά μας για το πρόγραμμα αυτό κοινωνικής αλλαγής και καινοτομία, για να μας παρουσιάσει την προφορική της ερώτηση. Παρακαλώ κυρία Στάινρικ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ναι πράγματι Είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που υιοθέτησε την αντιμετώπιση του θέματος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι τις επιστολές μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τις απάντησε, διότι υπήρχαν αρνητικές τοποθετήσεις συνεργατών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δική μας δουλειά μέσα στο ESCE. E. Και το ερώτημα είναι, το ζήτημα τώρα είναι το εξής. Η προφορική ερώτηση έχει κατατεθεί, είναι στη διάθεση του Επιτρόπου ή να την ξαναδιαβάσω για άλλη μια φορά για να την γνωρίσετε ποια είναι. Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, να σας δώσω το λόγο για να διαβάσετε το κείμενο, αλλά μπορώ να το κάνω κι εγώ. Εκτό αν οι συνάδελφοι κρίνουν ότι δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Κύριε Επίτροπε, γνωρίζετε λοιπόν την ερώτηση. Είναι η προφορική ερώτηση που σας υπευλήθη γραπτά βέβαια και για την οποία περιμένουμε να μας απαντήσετε. Ε, ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Πιστεύω ότι η απόφαση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν μια πολύ σημαντική απόφαση και γι' αυτό με ιδιαίτερη χαρά μπορώ να συζητήσω αυτό το θέμα μαζί σας σήμερα, ακόμα και αν υπάρχουν κάποια αντιφατικά, κάποιες αντιφάσεις γύρω από αυτό το θέμα. Πρώτον, να σας εξηγήσω τη χρονική συγκυρία για αυτή την απόφαση. Δύο κύριοι λόγοι υπάρχουν για την υιοθέτηση αυτής της απόφασης εφέτος. Πολιτικός λόγος ο πρώτος. Τον προηγούμενο τον Απρίλιο υιοθέτησε την ε, λήψη μέτρων και την προαναγγελία αυτής της απόφαση που θα γινόταν πριν από τα τέλη του έτους. Η επίσημη απόφαση 26 Νοεμβρίου και το περιεχόμενα και οι στόχοι ήταν γνωστοί από τον Απρίλιο. Είναι σημαντικό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γοργά να δράσει και να υλοποιήσει αυτά. Δεύτερον, λειτουργικά. Η απόφαση αυτή προβλέπεται ότι θα αρχίσει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2014 και αρκετοί πρέπει να προετοιμαστούν για τις αλλαγές που εισάγει και γι' αυτό έπρεπε να εγκριθεί επίσημα αρκετά νωρίς υπήρχε μια πιεστική ανάγκη από τα κράτη-μέλη ως προς αυτό, υπό αυτό το πρίσμα. Στην πρακτική εφαρμογή τρία παραδείγματα έχουμε ότι πρέπει αυτά όλα να γίνουν το 2013 να αναλυθούν δράσεις. Είναι τα εξής. Η εξέλιξη των κοινών ε, κριτηρίων ε, διαπίστευσης ε, και επιλογής όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών και τις επιλογές που θα γίνουν με βάση αυτά τα κριτήρια. Αναβάθμιση του καταλόγου υπηρεσιών στο εθνικό επίπεδο, ευθυγραμμιζόμενη με τον κατάλογο υπηρεσιών στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συναφή και συμπερίληψη των ιδιωτικών εταίρων σε αυτό το καθεστώς καταστατικό, ώστε να μπορέσουν τα κράτη-μέλη και οι φορείς να έχουν αρκετό χρόνο για να μπορέσουν να προετοιμαστούν να εμπλακούν και να είναι έτοιμοι και προετοιμασμένοι. Δεύτερο, όσον αφορά το θέμα της διακυβέρνησης ή διαχείρισης, το οποίο αναφέρθηκε σε προηγούμενη ανταλλαγή απόψεων ως θέμα, η λειτουργία της Γιούρες καθορίζεται από διάφορα νομοθετικά μέσα η δημιουργία, η στόχη και η ε, λειτουργία μέσω της διακυβέρνησης ε, από τον κανονισμό 492 του 2011 καθορίζεται για από το πλαίσιο περί δραστηριοτήτων εργαζομένων με βάση το άρθρο 46 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρηματοδότηση από τον Ιανουάριο 2014 θα διέπεται από τα οικονομικά, δημοσιονομικά μέσα, το ε, SCR e από τη μία πλευρά και το ESF από την άλλη και εθνικούς προϋπολογισμούς αφετέρου. Αντίθετα προς τα άλλα δύο τμήματα του τμήματος, ε, το μέσο για την ε, μακροχρηματοδότηση, η πρόσβαση, η προσπελασιμότητα στο EURES καθορίζεται και από ένα άλλο νομοθετικό μέσο, τον κανονισμό 492 του 2011 και γι' αυτό λοιπόν δεν είναι κάτι το αυθύπαρκτο ως ε, πρόσβαση για τη ρύθμιση της πρόσβασης, αλλά πρέπει να εξετάζεται πάντα σε συνδυασμό με αυτόν τον κανονισμό και σε συνάρτηση με αυτόν. Η απόφαση του Νοεμβρίου τι κάνει. Αποσαφηνίζει τα λειτουργικά μέσα και όργανα για την λειτουργικότητα αυτή, την, ε, ε, τις δράσεις των διαφόρων εμπλεκομένων, τους στόχους ε, και τον καθορισμό περί υπηρεσιών γενικότερα. Αυτοί οι κανονισμοί και διατάξεις βρίσκονται στο πλαίσιο του κανονισμού 4, του 2011. Μια νέα απόφαση δεν μπορεί να αλλάξει ούτε ουσιοδός τη δομή, τη διάθρωση, ούτε τη σύνθεση του δικτύου EURES. Εξ ου και αν η ίδια η συζήτηση αφορά τη διάθρωση του δικτύου Γιούρες και των δραστηριοτήτων του, αφορά πρώτα και κύρια τις διατάξεις για τον κανονισμό 492-2011 και όχι την ίδια την απόφαση αυτό τελώς. Η κύρια ε, τροποποίηση, οι κύριες τροποποίησεις που εισάγει αυτή η απόφαση είναι η εξής. Η αλλαγή ονόματος ή τίτλου όσον αφορά το σώμα αλλά η ε, σύνθεση και η λειτουργικότητα παραμένουν αναλύωτες. Δεύτερον, Όσον αφορά του ιδιωτικού εταίρους ε, για διάφορε δραστηριότητε, μπορούν να εντάσσονται σύμφωνα με εφαρμογή την ομολογία του ε, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, του 10. Η συμπερίληψη αυτών των νέων εταίρων είναι ένα άλλο επιχείρημα, ώστε νωρί να μπορέσει αυτή η απόφαση να ληφθεί και να λαμβάνεται, ώστε να μπορούν τα κράτη-μέλη και οι φορεί να προετοιμάσουν την ένταξή του στο δίκτυο και να μπορούν να λειτουργήσουν όπως πρέπει σωστά. Ένα άλλο, τρίτο σημείο, ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων διατηρείται και ενισχύεται, ώστε έτσι θα υπάρχει διαβούλευση για το πρόγραμμα δραστηριοτήτων σε σχέση με τα κράτη-μέλη, πράγμα που δεν συνέβαινε μέχρι σήμερα. Η διαφορά ποια είναι. Εργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τομείς σε σχέση με δραστηριότητες συμμετοχή σε δραστηριότητες όπως κατάρτιση, πληροφόρηση, ενημέρωση κτλ. Ωστόσο όμως από την άλλη πλευρά δεν θα συμμετέχουν για παράδειγμα σε συγκεκριμένα ε, το, θέματα και τομείς ε, όπως ε, για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που δεν θα είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν υπό όλες τις συγκυρίες σε τέτοιες δραστηριότητες. Στα θέματα όμως που θα είναι σημαντικά για αυτούς, οι εταίροι θα προσκαλούνται να συμμετάσχουν. Σας τα επιβεβαιώνω και επαληθεύω αυτά σήμερα και αν χρειάζεται θα μπορέσω να ενημερώσω σε σχέση με αυτά περαιτέρω αν χρειαστεί. Και εν τέλει, η αναθεώρηση του κανονισμού 492 του 2011 όσον αφορά το τμήμα του Γιούρες που προβλέφθηκε εξάλλου στο πρόγραμμα εργασίας για το 2013 ως στοιχείο αυτό θα γίνει υπό το άρθρο 46 της συνθήκης πάντα και γι' αυτό υπό την κανονική νομοθετική διαδικασία. Με άλλα λόγια τι σημαίνει αυτό. Οι ουσιώδει αλλαγέ για τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση του Γιούρε θα αποφασίζονται από του συνομοθέτε φυσικά πράγματι. Ελπίζω ότι έτσι μπόρεσα να αποσαφηνίσω κάποια πράγματα. Αν, μπορεί, αν πιστεύετε ότι θα ήταν επωφελέ, θα μπορούν οι υπηρεσίε να έχουν μια συνάντηση με του υπαλλήλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του ευρωβουλευτέ αρμόδιου για το χαρτοφυλάκιο επί του περιεχομένου αυτής της απόφασης για να δουν και να εξηγήσουν τι ακριβώς κάνει και τι δεν κάνει, ώστε να μπορέσουν να αποσαφινιστούν θέματα σε σχέση με την λειτουργία αυτής της απόφασης και την εφαρμογή της. Εν πάση περιπτώσει, στο τέλος τέλος ε, αυτής της διεργασίας, όταν θα έχει ε, προβεί ο συνομοθέτης σε έγκριση, θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει τις επιπτώσεις που μπορεί ίσως να υπάρχουν από αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Σέλφος Στάινμπρουκ, συνεχίζουμε. Κυρία Στάινμπρουκ, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε. Εδώ εμάς μας ενδιαφέρει κάτι που είναι θέμα αρχής ουσιαστικά. Η απόφαση εκτέλεσης ε, προβλέπει την κατανομή του Γιούρες σε EFSF και PC και για μας εξακολουθεί να ισχύει και ακόμα με την απάντησή σας η ασάφεια. Γιατί δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα των τριμερών διαλόγων σε σχέση με το ESF ε, και την άλλη συνιστόσα δεν την ανέμενε μια και αυτά θα αρχίσουν να ισχύουν από το 2014 ούτως ή άλλως. Και πρέπει να πω ότι μας περιγράψατε αυτά που από πλευρά τη εκτελεστικής απόφασης μπορούσαμε να διαβάσουμε οι ίδιοι, αλλά απουσιάζει πιστεύουμε εμείς η σαφήνεια στην τοποθέτηση για τα κομβικά σημεία τα οποία εμείς διατυπώσαμε στην ερώτησή μας. Μεταξύ της εκτελεστικής απόφασης αφενός και PSC βλέπω να υπάρχουν κάποιες εξαρτήσεις και θέματα τα οποία επηρεάζουν το ένα το άλλο στην αιτιολογική σκέψη της εκτελεστικής απόφασης αναφέρεται ότι μέτρα διασυνοριακά του Γιούρες μέσω του ESF θα χρηματοδοτούνται. Δεν το γνωρίζουμε όμως αυτό ακόμα και εσείς δεν το γνωρίζετε ακόμα εξαρτάται από τους τριμερείς διαλόγους μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου το τι θα γίνει. Δεν έχουν προχωρήσει τόσο πολύ ώστε εσείς να προδικάζετε κάτι τέτοιο. Προδικάσατε κάτι που εκκρεμεί ακόμα από την πολιτική απόφαση και δεν έχει καθοριστεί. Επίσης αναφέρεται ο νέος διαχωρισμός ESF και τα λοιπά και προβλέπεται και προδικάζεται ενώ αυτά δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα από πλευράς αποφάσεων. Εξάλλου και στο θέμα της για την κινητικότητα. Τι γίνεται. Και στα δύο κείμενα γίνονται αναφορές και καλύπτονται θέματα και για τους δείκτες αξιολόγησης. Για μένα είναι απόλυτα σαφές πλέον με αυτόν τον τρόπο ότι εσείς χωρίς να αναμείνετε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων που ευρίσκονται εν εξελίξη, τι κάνετε, δηλαδή προδικάσατε ποια θα είναι η πολιτική βούληση και σε ποιο αποτέλεσμα θα, θα καταλήγαμε. Αυτό δεν είναι νομίζω σωστό. Και αυτό εξ ονόματος των συνεισηγητών θα ήθελα να το αναφέρω. Είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι για αυτή την κατάσταση. Also, ε, Νομίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε σε ένα θέμα εδώ το οποίο είναι άκρος προβληματικό με αυτόν τον τρόπο. Απλά από το γραφείο της, τα γραφεία τους κάνουν πράγματα τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την πρακτική εφαρμογή, την καθημερινή πρακτική εφαρμογή. Τι λέει η πρακτική. Επί πολλά χρόνια, επί δεκαετίες ολόκληρες, είχαμε σημαντική βασικό θέμα για τις διαβουλεύσεις και όργανο για τις διαβουλεύσεις αυτές που χρηματοδοτούντουσαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Γιούρες. Οι διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις είναι αυτό το μέσο. Είναι ένα από τα πιο παλαιά μέσα όσον αφορά την ελευθερία κυκλοφορίας. Ανθρώπους που ζουν σε μια χώρα εργάζονται σε μια άλλη χώρα. Και ακριβώς σε αυτό το σημείο αναφύεται αυτό. Δεν αναφύεται ούτε στην Ισοκύπρο, ούτε στην Μάλτα, ούτε αλλού. Όμως στο κέντρο, στην καρδιά της Ευρώπης, σε πάρα πολλά σημεία αναφύεται και λειτουργεί έτσι. Και τι ήτανε τώρα, και σε σχέση με τις εκλογές για τις ε, εταιρικές σχέσεις ε, ήταν η βάση του κοινωνικού διαλόγου και λειτουργούσαν όλα με βάση τη συνθήκη. Με τον, τους παλαιούς κανονισμούς και διατάξεις του Γιούρες, οι κοινωνικοί εταίροι είχαν διαφορετικό ρόλο που διαδραμάτιζαν από τη νέα απόφαση που λαμβάνετε τώρα εσείς. Είχαν αυτοτελεί αυτόβουλο ρόλο, αυθύπαρτο ρόλο. Και είναι αυτονόητο ότι έτσι το Γιούρες όσον αφορά τον κανονισμό, οι διαβουλεύσεις ε, λειτουργούσαν σε σχέση με αυτές τις διασυνοριακές σχέσεις. Εσείς λέτε εντάξει, εντάσσονται πάλι. Αν δω το κείμενο, όχι, δεν εντάσσονται, ε, βρίσκονται εκτός. Λοιπόν, δεν είναι το αυτονόητο λοιπόν το οποίο ίσχυε μέχρι σήμερα Υπάρχει σημαντική υποβάθμιση και συρρήκνωση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων ακριβώς σε μια λειτουργία όπου είχαν αυξημένη σπουδαιότητα μέχρι σήμερα και όλο και μεγαλύτερη σημασία για μια ομάδα ανθρώπων. Και οι εργαζόμενοι ε, διασυνοριακά ήταν εκείνοι οι οποίοι αφορώνται άμεσα από αυτό. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, η ΕΣΕΦΕΣ και το, η άλλη συνιστός. Αυτά που λέτε είναι το μισό της αλήθειας. Δεν είναι η πλήρης αλήθεια δεν έχουμε καμία, κανένα σημείο αναφοράς, καμιά αναφορά στο ΕΣΕΦ γι' αυτό. Έχουμε κάποιες γενικές διατυπώσεις, γενικόλογα, όπου για κάποια εταιρική σχέση θα μπορούσαν κάποιοι να έκαναν αυτό το οποίο επιθυμούν. Ένα κράτος μέλος για παράδειγμα. Εδώ όμως κάνουμε λόγο για δύο ή τρία κράτη-μέλη ταυτόχρονα. Γιατί έχουμε την επιλογή μέσω αυτού του μέσου. Αν θα έχει το κράτος μέλος από πλευρά του τέτοιες προτεραιότητες για τις επενδύσεις. Αν δεν έχει τέτοιες προτεραιότητες δεν θα γίνονται αυτές οι δράσεις. Προέρχομαι από μια τέτοια περιοχή όπου έχουμε την Πολωνία, την Σιεχία και την Γερμανία. Αν μία από αυτές τις χώρες δεν, θέλουν, δεν θέλει αυτές τις ε, προτεραιότητες, δεν θα υπάρχουν κονδύλια. Είναι απόλυτα ανόητο, παράλογο να έχουμε εθνικό πρόγραμμα το οποίο θα εξαρτάται από την εθνική υλοποίηση και εκτέλεση για να χρηματοδοτηθεί κάτι το οποίο είναι ευρωπαϊκού χαρακτήρα, ευρωπαϊκής διάστασης. Μόνο ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πρέπει και μπορεί να διασφαλίζεται. Μετά, στον κανονισμό έχετε κάτι εκείνοι οι οποίοι θα παίρνουν αυτά τα κονδύλια πρέπει να έχουν και κάποιες επιδόσεις, να δίνουν κάποιο αντίτιμο. Σε αυτόν τον κατάλογο όμως ε, επιδόσεων δεν αναφέρονται οι κοινωνικοί εταίροι. Υπάρχουν ε, υπηρεσίες ή δράσεις που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε που δεν υπήρχαν πριν. Υπάρχει δεσμευτικός χαρακτήρας λοιπόν που καθιστά ανέφικτη τη χρηματοδότηση των εταίρων μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Γίνεται λόγος και για υπηρεσίες που πρέπει να ε, παρέχονται και μάλιστα με υποχρεωτικό χαρακτήρα στον κατάλογο που και αυτές πάλι δεν μπορούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο να, γίνεται, να γίνονται. Αν είναι υποχρεωτικά όλα αυτά, τότε αν δεν ε, υλοποιούνται αυτές οι υποχρεώσεις δεν θα δίνονται κονδύλια στους εταίρους. Επί δεκαετίες ένας επιτυχής θεσμός που λειτουργούσε υπέρ των Ευρωπαίων εργαζομένων, εδώ συρρυκνώνεται ας το πω έτσι, ε, καταλήγει σε μια ελεηνή κατάσταση. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα με τη νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Απευθύνω έκκληση σε εσά αυτό το σφάλμα αμέσω να το επανορθώσετε και να αναλάβετε τα αναγκαία βήματα και διαβήματα με το Κοινοβούλιο να επανορθωθούν τα πράγματα. Εμείς έχουμε πείρα με τις στενές επαφές ε, και τη στενή σχέση με τους εταίρους στις διασυνοριακέ σχέσει. Δεν πρόκειται εδώ για τεράστια κονδύλια. Πρόκειται για ένα σημαντικό πλαίσιο διαρθρωτικό με μικρά κονδύλια που απαιτούνται που έχουν όμως τεράστια σπουδαιότητα. Αν δεν γίνει αυτό θα κάνουμε τεράστιο σφάλμα για το μέλλον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Παρ' όλα αυτά θέλω να προσυπογράψω τις γενικές τους ιδέες και αυτά που είπε η συγγητριά μας ε, σχετικά με το ε, ΨΥ ε, και για τις διασυνοριακές σχέσεις, γιατί στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου έχουμε αναλάβει να ενισχύσουμε αυτές τις διαδικασίες. Θα ήθελα, θα ήθελα να επανέλθω ε, στην πρόταση για ε, ε, τροποποίηση του πόρταλ του Γιούρες. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει δυνατότητα πληροφόρησης Ε, νομίζω λοιπόν λέω ότι θα πρέπει ε, οπωσδήποτε να είμαστε σίγουροι ότι δεν κάνουμε, δεν βάζουμε κυβάκια έτσι κομματάκια σε ένα παζλ και ότι θα πρέπει να βρεθούν ε, κάποιες αξιόπιστες μέθοδοι πρόσβασης στην εργασία έστω και αν το αρχικό προφίλ του ετούντος εργασία δεν είναι ακριβώς αυτό που θα τέριαζε εξ αρχής. Επίσης η πρόταση της Κομισιόν Νομίζω ότι αυτή, αυτή η πρόταση για τις ε, σχέσεις ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Συντονιστικό Γραφείο και τον ε, ε, συντονισμό του Γιούρες. Δεν καταλαβαίνω πολύ καλά αυτά τα προφίλ και πώς αντιστοιχούν. Εγώ μερικές φορές βλέπω ότι είναι κοινέ οι αρμοδιότητες, άρα θα υπήρχε επικάλυψη. Τέλος να πω ότι στα πλαίσια του τριμερού διαλόγου, ε, που είναι ο πρώτος στον οποίο προσωπικά συμμετέχω και επομένως ε, δεν έχω έτσι την αρχαιότητα κάποιων συναδέλφων, όμως βλέπω ότι δύσκολα μπορούμε να δεχτούμε στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων να μας ανακοινωθεί ότι τροποποιεί η Κομισιόν το ΕΡΕΣΑ και προτείνει, το Γιούρες και προτείνει διαφορετική χρηματοδότηση λαμβάνοντας ε, υπόψη στοιχεία τα οποία ουδόλως είχαμε ε, στη διάθεσή μας. Τώρα μας λένε ότι το Eures θα κοστίσει περισσότερο, αλλά επί τη βάση του νέου σχεδίου βέβαια. Αλλά δεν, έχουν, δεν είχαμε εμείς στη διάθεσή μας το σχέδιο αυτό. Ε, και επομένως εγώ θα συμφωνήσω απολύτως με αυτά που λέει η κυρία Στάινρουκ και πιστεύω ότι θα έπρεπε είτε να μας παρουσιαστεί, να μας υποβληθεί το σχέδιο πριν, είτε πολύ αργότερα. Όμως με καμία περίπτωση στη διάρκεια της ε, διαπραγμάτευσης. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, κυρία Πρόεδρε, δεν κατάλαβα. Θα είμαι πολύ σύντομη, κύριε Επίτροπε. Εδώ επιτρέψτε μου να σας διαβάσω ένα νομικό κείμενο γι' αυτό. Εντάξει, δεν είναι ότι το καταλαβαίνω, θα κάνω, πώ το καταλαβαίνω. Κάποια μπορώ να τα παρακολουθήσω, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ περίπλοκο και αυτό ακριβώ είναι το δύσκολο εδώ, ότι είναι ασαφέ το θέμα. Συμφωνώ με αυτά που είπαν οι συναδελφοί, ότι την ανταλλαγή αυτή απόψε έπρεπε να την είχαμε νωρίτερα. Τώρα βρισκόμαστε εν μέσω ενό τριμερού διαλόγου, δεν έχουμε στήριξη από το Συμβούλιο, δεν έχουμε πληροφορίε, δεν έχουμε τίποτα. Είμαστε μπροστά σε ένα τείχος και επειδή δεν υπήρξε καμιά ένδειξη από την Επιτροπή όσον αφορά το περιεχόμενο κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου, δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε. Εσείς λέτε ότι αυτό δεν επηρεάζει τα δημοσιονομικά. Για μας όμως δεν μπορούμε να το ξέρουμε τώρα στη μέση του τριμερούς διαλόγου. Είναι δηλαδή σαν να προσπαθούμε να αλλάξουμε τα πράγματα στη μέση της διαδρομής. Θα ήθελα λοιπόν έχω περισσότερες πληροφορίες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μια λύση πρέπει να βρεθεί στο πρόβλημα. Και η... συμφωνώ με την εισηγήτρια και εγώ για όλα όσα είπε. Πρόεδρος. Από μου εγώ θέλω να πω στον ε, Επίτροπο, αλλά το είπα και στον κύριο Ρισελιέ με τον οποίο μίλησα, ότι καταλαβαίνω πως ε, υπάρχει ένα θέμα με το πακέτο για την απασχόληση. Αλλά εσείς μιλάτε, λέτε ότι 1η Ιανουαρίου 2014 είναι η ημερομηνία θέση ισχύ. Ναι, αλλά η μεταρρύθμιση του Γιούρες είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση και δεν νομίζω ότι η μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Ταμείου, τη τομή Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, ε, της βοήθειας για τους πιο ευάλωτους και μπορεί να ξεχνάω κι άλλα, είναι λιγότερο σημαντικά από πλευράς ε, ανάγκης διοικητικής προσαρμογής. Συνεπώς, γιατί λέτε ότι αυτό ήταν πιο επίγον από τα άλλα, στο οποίο επίσης έχουμε συναπόφαση. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Μας δημιουργεί πρόβλημα χρονοδιαγράμματος, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η συνθήκη της Λισαβόνας. Σας παρακαλώ να μας απαντήσετε. Και να πω ήδη από τώρα στους συναδέρφους ότι Μόλις φύγει ο Επίτροπος, ξεκινάμε συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε με αυτό. Ε. Ο Επίτροπος. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση αυτή και ολόκληρη υπόθεση. Εμείς προσπαθούμε να προσφέρουμε ό,τι στοιχεία έχουμε, και εγώ και το προσωπικό μας. Θέλουμε έγκαιρα να σας εξηγήσουμε τις προτάσεις μας και ειλικρινά λυπάμαι που επειδή έπρεπε να αξιολογήσουμε όλες τις πτυχές, κάποιες από τις απαντήσεις μας έφτασαν σε εσά πολύ αργά. Θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Αυτό είναι το ιστορικό, αυτή είναι η ιστορία από πίσω. την η εξήγηση των όσων ανέφερε η κυρία Στάινρουκ. Εν πάση περιπτώσει. Πιστεύω ότι εδώ υπάρχουν διάφορες σημαντικές πτυχές που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Όταν ε, μιλάμε για μια υπηρεσία, το εννοούμε. Ε, λαμβάνουμε υπόψη μας την ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι πραγματικά τραγική και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε μιλήσει ξανά και ξανά για αυτό το θέμα. Όταν επισκέφθηκα χώρες ε, μέλη πρόσφατα, τι με ρωτούσε ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι. Μου λέγανε, μα η Επιτροπή τι θέλει τελικά, να σηκωθούν να φύγουν οι νέοι από τις χώρες τους, να μεταναστεύσουν. Η απάντησή μου είναι ότι η Επιτροπή θέλει οι άνθρωποι αυτοί να βρουν δουλειές και να βρουν δουλειά εκεί που υπάρχει δουλειά. Όλο και περισσότερο εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης και των επιπτώσεών της, απασχόληση θα υπάρχει στο εξωτερικό. Και θα υπάρχει απασχόληση εφόσον υπάρξει καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Και υπογραμμίζω και πάλι, είναι επίγον το θέμα, όντως, επίγει το θέμα της απασχόλησης, γι' αυτό έχουμε και το πακέτο για την απασχόληση και η απόφαση που συζητάμε τώρα υπογραμμίστηκε την άνοιξη στο πακέτο για την απασχόληση. Και έτυχε και θετική υποδοχή στο εγγραφό αυτό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορείτε να το αρνηθείτε αυτό. Όσον αφορά τώρα τη λειτουργία του Γιούρες, εδώ νομίζω ότι υπάρχει ένα ισχυρό επιχείρημα να αναλυφθεί δράση. Έχετε δίκιο σε αυτό. Ακόμα και αν η δράση σημαίνει προετοιμασία για κάτι το οποίο θα πάρει χρόνο να τεθεί και σε εφαρμογή. Όσον αφορά την σχέση ανάμεσα στη λειτουργία του γύρους από τη μία και τη μελλοντική του χρηματοδότηση από την άλλη, εδώ πρέπει να δούμε χρονικά πώς έχει το πράγμα. Γιατί εμεί θέλουμε βέβαια να βελτιωθεί η λειτουργία ενός συστήματος, ενός μέσου που έχουμε ήδη, που έχει τεθεί σε εφαρμογή και που πρέπει να ανταποκρίνθει στην τρέχουσα κατάσταση. Από την άλλη μεριά μιλάμε για το μελλοντικό προϋπολογισμό Ό,τι και αν λέμε για το πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και καινοτομία έχει να κάνει με την περίοδο 2014 με 2020. Και πολλές φορές μέχρι τώρα έχουμε πει, και το επαναλαμβάνω και τώρα, ότι εάν συνεχιστεί η συζήτηση για το πρόγραμμα αυτό, ίσως θα έχουμε και νέα στοιχεία για το EURES. Και εφόσον συμβεί αυτό, εννοείται ότι θα ανταλάβουμε λάβουμε υπόψη μας. Είτε στα πλαίσια της αναθεώρησης του κανονισμού, που σας είπα στην ε, αρχή εισαγωγικά, ή ακόμα και αργότερα, αν αυτό αιτιολογείται. Ακριβώς επειδή είμαστε σε μια κατάσταση όπου επήγει να προχωρήσουμε. Θέλουμε να έχουμε δίπλα μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους κοινωνικούς εταίρους. Γνωρίζουμε ποιες είναι οι ευθύνε μας. Ότι οι κοινωνικοί εταίροι δηλαδή πρέπει να συμμετέχουν και να διαβουλευόμαστε μαζί τους για κάθε απόφαση που παίρνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την πολιτική μας. Και έτσι η απόφαση του Νοεμβρίου πιστεύουμε εμείς ότι δεν επηρεάζει καθόλου αρνητικά τον ρόλο που παίζουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Τώρα υπάρχουν και κάποια τεχνικά ζητήματα. Η η κατάσταση απαιτεί παρετέρω συζήτηση και προβληματισμό. Γι' αυτό ήθελα να τα διευκρινίσω όλα αυτά. Και αυτά που είπατε για την επαγγελματική κατάρτιση και το ρόλο των κοινωνικών εταίρων γενικά. Γνωρίζω επίσης ότι ακόμη και σας είναι λεπτομερή απάντηση, δεν σημαίνει ότι έτσι κλείνει και η συζήτηση. Αν μη τι άλλο υπάρχουν και δημοσιονομικές πτυχές, άρα η συζήτηση πάνω σε αυτές θα συνεχιστεί. Όχι μόνο στο Κοινοβούλιο αλλά και στο Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα προσβλέπω σε παρετέρω συνεργασία μεταξύ μας και εφόσον το επιθυμείτε και είναι αναγκαίο, ευχαρίστω να σας απαντήσω και γραπτά. Είμαστε στους κανόνες της Λισαβόνα. Αυτούς ακολουθούμε. Και ξέρουμε ποιε είναι οι υποχρεώσει μας. Δεν τις ε, αρνούμαστε και ούτε θα κάνουμε καμία εξαίρεση σε αυτές. Πρόεδρος, κύριε Επίτροπε, ξέρω ότι έχετε πολλή δουλειά, οπότε σας ευχαριστούμε που ήρθατε για να απαντήσετε σε αυτή την προφορική ερώτηση για ένα θέμα που είναι τόσο πολιτικό όσο και νομικό. Αλληλογραφούμε εδώ και καιρό. Η πρώτη επιστολή που σας στείλαμε εκ μέρους των συναδέρφων ήταν στις 4 Ιουλίου του 2012. Η ανταλλαγή που είχαμε είχε να κάνει περισσότερο με την πολιτική διάσταση της μεταρρύθμισης που επιθυμείτε. Παραμένει το νομικό. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που ήρθατε και για τόσα μας είπατε μέχρι τώρα. Δίνουμε ραντεβού του χρόνου, ε. Ευχαριστώ και τους ε, συναδέρφους. Φροντίστε τώρα να έχουμε για λίγο και κλεισμένο των θηρών συνεδρίαση για να αποφασίσουμε μεταξύ μας τι συνέχεια θα δώσουμε σε αυτή την υπόθεση. Αυτό σημαίνει ότι οι παρατηρητές παρακαλώ να βγουν από την αίθουσα, οι εκπρόσωποι της Επιτροπής επίση, οι επισκέπτες. Εδώ θέλω να μείνουν μόνο τα μέλη της Επιτροπής μας, η νομική υπηρεσία, οι συνεργάτες και οι πολιτικοί υπάλληλοι. Ευχαριστώ. προφορική τροπολογία που έχει υποβάλει η ομάδα του ΕΛΚΕ, η οποία ζητάει την φράση διασφαλίζοντας ε, ε, διασφαλίζοντας το μέλλον των, πολιτών, των νέων πολιτών της Ευρώπης ή νομίμως διαμενόντων. Και έχουμε και μία δεύτερη προφορική τροπολογία από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες μέχρι την ηλικία των 25 ετών ε, και σε περίπτωση διπλωματούχων μέχρι την ηλικία των 30. Δεν ε, ε, υπάρχει, βλέπω, καμία αντίθεση. Επομένως, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ο συμβολός Α. Οι άλλες τροπολογίες καταπίπτουν. Και μετά την παράγραφο 2 έχουμε την τροπολογία 18 της κυρίας Άμιλη Τουρίνεν. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 19 έχει αποσυρθεί. Μετά την παράγραφο αυτή υπάρχει η τροπολογία 20 η οποία έχει καλυφθεί. Και μετά την παράγραφο 2 έχουμε και την τροπολογία 21 Αλεξάνδρ Σέρκας. Υπέρ κατά αποχές ε, θα δούμε. Ε, λοιπόν, ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 21. Le vote est ouvert, tout le monde a pu voter le vote. Άρχεται η ψηφοφορία, ψήφισαν όλοι, πέρασε. 18 υπέρ, 13 κατά, 4 αποχές, επομένως εγκρίνεται. Τροπολογία 22 του ιδίου, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 ορία έχει αποσυρθεί. Ψηφίζουμε λοιπόν μετά την παραγραφό 2 το συμβιβασμό Β που έχει παρουσιαστεί από τρεις ε, ομάδες με προφορική τροπολογία των φιλελευθέρων. Δεν υπάρχει αντίθεση όσον αφορά την προφορική τροπολογία. Όχι, ψηφίζουμε το Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 2 τροπολογία 25 Αλεξάνδρος Έρκας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 του ιδίου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παραγραφό 2 οι τροπολογίες 27 και 28 καταπίπτουν. Ψηφίζουμε την τροπολογία 29 τζάμπα όρη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3 νέα. η ε, επόμενη τροπολογία, Έμιλη Τουρινέν υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικέ σκέψεις Α, τροπολογία 2, Αλεξάνδρου Σέρκας, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Β, τροπολογία 3, Μιλακαμπνόχ, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4, Αλεξάνδρου Σέρκας, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 ε, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η Αιτιολογική σκέψη Β νέο, τροπολογία 6 έχει αποσυρθεί. Ε, τροπολογία 7 Αλεξάνδρο Σέρκα ε, για την επόμενη αιτιολογική σκέψη υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται μετά το σε τροπολογία 8 Έμιλι Τουρίνεν υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 9 ε, Αλεξάνδρο Σέρκα υπέρ κατά. Ποιο είναι υπέρ? Contre. Υπέρ κατά. Αποχές. Νομίζω ότι θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση παρόλα αυτά. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί, θα δούμε. Ψήφισαν όλοι, πέρας. 17 υπέρ, 12 ε, κατά, 5 αποχές, επομένως όντως εγκρίθηκε. Μετά το C, τροπολογία 10, Αλεξάνδρο Σέρκα με την προφορική τροπολογία που έχουν υποβάλει οι πράσινοι. Δεν υπάρχει πρόβλημα με την τροπολογία αυτή. Επομένω, ψηφίζουμε την τροποποιημένη τροπολογία υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Μετά το ΔΕΛΤΑ τροπολογία 11, Τζαμπαωρή, με προφορική τροπολογία. Δεν υπάρχει αντίθεση σε αυτή την προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροποποιημένη τροπολογία υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Όσον αφορά τα σημεία, η τροπολογία έρκαση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σύνολο του κειμένου ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Ε, ψήφισαν 36, 34 υπέρ, μία ψήφος κατά, μία αποχή. Nous en venons nous, à notre ordre du jour que nous reprenons au point. Ξαναρχίζουμε λοιπόν την ημερήσια διάταξη. Την είχαμε αφήσει στο σημείο 4 και θα δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Καπνόρ, ο οποίος ε, θα πάρει τη θέση της κυρίας Μακιντάιερ. για την εξέταση των 46 τροπολογιών όσον αφορά την ε, ε, γνωμοδότηση για τη διακυβέρνηση της ενέας αγοράς. Είναι γνωμοδότηση για θέμα που είναι η ΙΜΚΟ αρμόδια επί της ουσίας. Ε, κύριε Καπνόχα, έχετε το λόγο. Ladies Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους της κυρίας Μάκιντάιρ μιλάω η οποία δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, εκ μέρους της, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι υπέβαλαν τροπολογίες στην γνωμοδότηση αυτή. Η συγκέντριά μας μπορεί να υποστηρίξει τις περισσότερες από τις ε, υποβεβλημένες τροπολογίες. Κάποιες όμως από αυτές δεν μπορεί να τις στηρίξει. Κάποιες από τις τροπολογίες σίγουρα φέρνουν νέες ιδέες και συνεισφέρουν προκειμένου η γνωμοδότηση αυτή να βελτιωθεί. Η συγκήτρια ελπίζει ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και να καταλήξουμε σε μια πολύ καλή γνωμοδότηση με σαφείς συγκεκριμένες προτάσεις για την υπεύθυνη επί της και αρμόδια επί της επιτροπή. Θα προτείνω μάλιστα και συμβιβαστικές τροπολογίες και θα έρθει και σε επαφή με συναδέρφους που έχουν υποβάλει τροπολογίες για περιπτώσεις δηλαδή όπου θα ζητήσει διευκρινήσεις και ενδεχομένως θα υποβάλει προφορικές τροπολογίες. Πιστεύει πάντως η συγκήτρια ότι δεν πρέπει να υπάρξει επικάλυψη με την δουλειά που κάνει η ΙΜΚΟ, που είναι η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, και ότι πρέπει να σταθούμε στις αρμοδιότητες της δικιάς μας Επιτροπής όσον αφορά την ενιαία αγορά. Τα κύρια σημεία τώρα που θέλω να υπογραμμίσω είναι τα εξή. Η ενιαία αγορά είναι κάτι που πάντα πιστεύαμε ότι έχει έναν ρόλο κλειδί να παίξει προκειμένου να πετύχει η στρατογική για το 2020 να ενισχυθεί η βιώσιμη ανάπτυξη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής σημειώνεται ότι προκειμένου να επιτευθούν οι στόχοι της στρατηγικής μας για το 2020, πρέπει να εφαρμόζεται καλά η κοινοτική νομοθεσία. Και σημειώνει ότι υπάρχουν πάρα πολλές οδηγίες οι οποίες δεν έχουν ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία έγκαιρα και ότι διαπιστώνεται ότι οι οδηγίες αυτές είναι όλο και περισσότερες όπου η ενσωμάτωσή τους δηλαδή στην εθνική ε, διαδικασία γίνεται μετά τη λήξη της προθεσμίας ή μάλιστα μετά από προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και ότι πολλές φορές δεν εφαρμόζονται και στην πράξη ικανοποιητικά. Η γνωμοδότηση λοιπόν θέλει να αντιμετωπίσει τέτοιες ε, περιπτώσεις και να δει πώς μπορούν να γίνουν ε, βελτιώσεις για να διασφαλιστεί η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, η καινοτομία και η οικονομική ανάπτυξη να μειωθεί το διοικητικό άχθος, για παράδειγμα, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μικροεπιχειρήσεις. Επίσης, η ιδέα του να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας, ένα ενιαίο γκισέ, όπως το λέμε, που να μπορεί να απευθυνθεί κανείς για να τακτοποιήσει τα γραφειοκρατικά του ζητήματα. Επίσης, πόσο μεγάλη σημασία έχει και η αξιολόγηση της νομοθεσίας για να έχουμε μια καλύτερη νομοθεσία μέσα στα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Τα επόμενα δύο χρόνια μάλιστα. Παρακαλώ, κύριο Στέρκα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εκ μέρου ε, του συναδέλφου Κοτσολίνου που δεν είναι εδώ σήμερα, να ευχαριστήσω την κυρία Μάκιντάιρ για την δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Και θέλω να υπογραμμίσω δύο στοιχεία συγκεκριμένα, τα οποία μπορεί να είναι αποφασιστική σημασία για την ε, θέση που θα υιοθετήσουν οι σοσιαλιστέ στο μέλλον. Και θα αναφερθώ σε μια πολύ συγκεκριμένη τροπολογία, αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση και η δεύτερη θα είναι πιο γενική. Ο κύριο Γκαμπνό μας ε, είπε ότι θα ληφθούν υπόψη διάφορε τροπολογίες. Η πρώτη τροπολογία που πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντική, τρεις βασικά, είναι η 31, η 32 και η 33 της κυρίας Στάινερ, του κυρίου Χιούς και δικιά μου. Υπάρχει εδώ ένα στοιχείο που πιστεύουμε ότι είναι ζωτική σημασία. Καλύτερη νομοθεσία, να νομοθετούμε καλύτερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να νομοθετούμε πια και τα κοινωνικά ζητήματα. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι ακούγεται ιδέα ότι για να μην δυσκολευόμαστε στην νομοθέτηση κάποιων δύσκολων μέτρων, ας μην νομοθετούμε καθόλου. Ε, δεν είναι σωστό αυτό. Στην δεύτερη παράγραφο λοιπόν δεν πρέπει να λέει αυτό που λέει τώρα ότι ιδιαίτερα σε θέματα απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων δεν πρέπει να λέγεται αυτό. Δεν μπορεί να λέμε ότι στο δομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων υπάρχουν μειονεκτήματα, προκειμένου δηλαδή να έχουμε μια καλή νομοθεσία. Για μας αυτό είναι απαράδεκτο για μας τους σοσιαλιστές. Γιατί συνέχεια μιλάμε για διοικητικά εμπόδια κάθε φορά που θέλουμε νομοθεσία για τα κοινωνικά δικαιώματα. Υπάρχει και μια άλλη που τουλάχιστον από τα αγγλικά που γνωρίζω εγώ δεν το καταλαβαίνω. Αυτό το καινούριο, το να θέλουμε άλλο κανόνα για αυτούς που είναι μέσα και άλλος για αυτούς που είναι έξω, δεν καταλαβαίνω. Τι σημαίνει αυτό, ότι κάθε νέα διάταξη θα καταργεί οποιαδήποτε προηγούμενη διάταξη όσο καλή και αν είναι αυτή, έτσι αυτόματα. Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο οι διατάξεις πρέπει να αξιολογούνται ανάλογα με την αξία τους. Το να λέμε ότι κάθε νέα διάταξη εξαφανίζει τις προηγούμενες, ακόμη και αν δεν είναι τις ίδιες ακριβώς φύσεις, δεν είναι σωστό. Αυτή λοιπόν η παράγραφος 8 δεν μας αρέσει, γι' αυτό και θέλουμε να διαγραφεί. Αν τώρα αναλύσετε και την τροπολογία 7, θα καταλάβετε τι πιστεύουμε εμείς για αυτή την υπόθεση. Είναι του κύριου Κοτσολίνο. Έτσι. Η ενή αγορά είναι πολύ σημαντική, δεν υπάρχει αμφιβολία. Παίζει επίσης έναν ρόλο αποφασιστική σημασία για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το πρόγραμμα για την Ευρώπη του 2020. Έχει να παίξει, λέμε, σημαντικό ρόλο. Αλλά δεν είναι το μόνο. Εμείς πιστεύουμε πιστεύουμε ότι η εσωτερική αγορά θα βελτιώσει και την απασχόληση και την ευημερία των πολιτών μας. Δεν είναι οι πολίτες που πρέπει να εξυπηρετούν την αγορά, αλλά η αγορά να εξυπηρετεί τους πολίτες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ζητάει άλλο το λόγο. Παρακαλώ κύριε Κόζα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, θα είμαι μάλλον σύντομος. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εργασία που έχει κάνει. Συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρξουν ε, συμβιβαστικές ε, λύσεις, γιατί ε, υπάρχουν και τροπολογίες οι οποίες δίνουν τελείως διαφορετικές ε, θέσεις. Πάντως πρέπει να πούμε ότι οι παρούσες ε, λύσεις δεν οδηγούν σε πλήρη αποτελέσματα. Χρειάζονται περαιτέρω μέτρα έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η ενιαία αγορά. Όμως η θέση κάποιων μερών δεν είναι η κατάλληλη. Επομένως πρέπει να φτάσουμε σε συμβιβαστικές λύσεις. Όταν μιλάμε για κρατικά μονοπόλια, ας πούμε, όταν μιλάμε για την ε, ε, συμφιλίωση διαφόρων ε, συμφερόντων κλπ. Είναι απαραίτητο όλες οι πολιτικές ομάδες να δουν κάποιες θέσεις και αν είναι δυνατόν να τις συμφωνήσουν από κοινού. Τέλος, να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να εγκριθούν διαφορετικά μέτρα για τους αναπήρους, για τους ανθρώπους με ειδικέ ανάγκες. Εγώ θα ήθελα να έχουμε περαιτέρω συνεργασία και με την εισηγήτρια έτσι ώστε να πετύχουμε και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την συγγήτρια για την έκθεσή της που αποτελεί μια πολύ καλή βάση εργασίας. Έχουμε υποβάλει ε, ως φιλελεύθεροι κάποιες τροπολογίες. Όντως υπάρχει το ζήτημα αυτό για την ανεργία των νέων. Ε, χρειαζόμαστε θέσεις εργασίας για αυτούς τους ε, νέους και βεβαίως ε, αυτές ε, οι θέσεις εργασίας μπορούν να δημιουργηθούν στα πλαίσια των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Άρα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα βελτιστοποίησης και μεγιστοποίησης των επιχειρηματικών ευκαιριών στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλα αυτά συνάδουν με την σωστή υλοποίηση και ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Είναι προφανές ότι μόνο αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις θέσεις και επομένως πρέπει προς αυτήν την κατεύθυνση να ε, εργαστούμε. Είμαι πεπισμένη ότι τελικά σε καλή συνεργασία και με την εισηγήτρια θα φτάσουμε σε μία έκθεση η οποία ε, θα ε, ανταποκρίνεται στις συζητήσεις που είχαμε. Κύριε Κομπνόχ, θέλετε να πάρετε το λόγο να ολοκληρώσετε. Ε, όχι, θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω για τη συζήτηση, να ευχαριστήσω όσους παρενέβησαν ε, και σας ευχαριστώ πολύ. Άψογα, λέει η Πρόεδρος. Επομένως, ε, επομένως έχουμε συμβαστικές τροπολογίες. Donc nous voterons le 14... Θα ψηφίσουμε τη 14η ε, Ιανουαρίου, ενώ η ΙΜΚΟ θα αποφασίσει 23-24 Ιανουαρίου, τότε που έχουν δηλαδή την δικιά του συνάντηση. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη θα φτάσουμε στο σημείο 9, το οποίο αφορά τον αντίκτυπο τη οικονομικής κρίσης στην ισότητα των φύλων και στα δικαιώματα της γυναίκας. Πρόκειται για έκθεση πρωτοβουλίας επί του οποίου η συνάδελφος Γκαμπριέλ ε, Τσίμερ ε, θα αντικατασταθεί από τον συνάδελφο Τσίμερ. Και πρόκειται για... Ε, από τον κύριο Χέντελ, συγγνώμη. Έχετε το λόγο. κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος κυρία Τζίμερ που δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ. Βεβαίως ε, μου έχει στείλει την θέση της έτσι ώστε να σας την υποβάλω. Σας ε, θυμίζω ότι η κυρία Τσίμερ έχει υποβάλει ψήφισμα ενώπιον της Επιτροπής για την ισότητα ε, των ανδρών και των γυναικών στην εργασία. Λυπούμεθα γιατί μέχρι τώρα η Κομισιόν δεν έχει απαντήσει στις αποφάσεις του Κοινοβουλίου του 10 και του 11 και καμία νομοθετική πρωτοβουλία δεν έχει ληφθεί κατά αυτή την έννοια η προσπάθεια επίτευξης ισότητας ανδρών και γυναικών στην πολιτική απασχόλησης αποτελεί για μία ακόμα φορά ε, προτεραιότητά μας. Ε, με το παρόν πρόγραμμα και λόγω ακριβώς της παρούσης καταστάσεως κρίσεως την οποία διανύουν οι περισσότερες ε, χώρες διαπιστώνουμε ότι οι πολίτες πλήγονται, πλήττονται από την κρίση διαφορετικές στιγμές και με διαφορετικούς τρόπους. Το 2009 είχαμε 9,1 ε, ε, νεανική ανεργία και 9,2 στις γυναίκες. Ε, μετά είχαμε την κρίση και η τάση οδηγεί, η τάση ήταν να είναι περίπου ίδιο το ποσοστό ανεργίας ανδρών και γυναικών το 2011. Η ανεργία ήταν 9,7 στις γυναίκες, 9, διορθώνω, 9,7 στους άντρες και 9,8 στις γυναίκες. Όμως, ε, διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν μεγάλες περικοπές στο δημόσιο τομέα, άρα επλήγονται ε, περισσότερο οι γυναίκες. Αυτή τη στιγμή 70% ε, των ε, ε, δημοσίων θέσεων εργασίας καλύπτονται από γυναίκες ε, στην Ελλάδα, οι κοινωνικές περικοπές, οι περικοπές στην εκπαίδευση και στο δημόσιο τομέα γενικότερα, εκεί όπου δηλαδή είναι περισσότερες οι γυναίκες, οι περικοπές αυτές ήταν πάρα πολύ μεγάλες και έπληξαν τις γυναίκες περικοπές έχουμε και σε όλες περίπου τις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, και επομένως αυτά τα μέτρα τελικά καταβαραθρώνουν την κατάσταση σε αντίθεση με όλες τις προσπάθειες που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και αντίθετα με τις περιαντιθέτου δηλώσεις μας ότι δηλαδή θέλουμε να χτυπήσουμε την ανεργία και κυρίως την ανεργία των γυναικών. Βλέπουμε ότι οι γυναίκες έχουν πάντα μεγαλύτερη ανεργία από ότι οι ε, ε, άνδρες. Αλλά τούτη τη στιγμή η διεξασφάλιση θέση εργασίας είναι και η εξασφάλιση της μη κοινωνικής περιθεριοποίησης. Ε, οι γυναίκες, ειδικά οι γυναίκες με αναπηρία, βεβαίως είναι ιδιαίτερα ευάλωτες, λαμβάνοντας υπόψη ότι ε, τα άτομα με αναπηρία γενικότερα παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό Nicht alle Λοιπόν, λαμβάνοντα υπόψη ότι ε, οι ανάπηροι είναι περισσότερο ευάλωτοι, καταλαβαίνουμε ότι οι γυναίκε ανάπηρε είναι ακόμα πιο ε, ευάλωτε. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Θα θέλαμε ε, στο επόμενο FSE τα ερωτήματα αυτού του είδους και τα ζητήματα αυτού του είδους να ληφθούν υπόψη έτσι ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θα πρέπει να υπάρξει και όσον αφορά την απασχόληση αλλά και γενικότερα τα κοινωνικά ζητήματα θα πρέπει να υπάρχει λέγω ισότητα μεταξύ ε, των ανδρών και γυναικών. Θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια πραγματικής συμφιλίωσης τη επαγγελματική ζωή με την οικογενειακή ζωή που και αυτή πλήττει περισσότερο τι γυναίκε θα πρέπει να υλοποιηθούν μέτρα τα οποία θα ενθαρρύνουν τους άνδρες ε, να πάρουν ε, γονεϊκή ε, άδεια και να ασχολούνται περισσότερο με τις οικογένειές τους. Οι μελέτες και οι αναλύσεις όσον αφορά την ε, μεγάλη παρουσία των γυναικών ε, στα ποσοστά φτωχών ε, ανθρώπων μας οδηγεί στο συμπέρασμα στην ανάγκη περισσότερο να προχωρήσουμε στους, σε κανόνες για την ισότητα των μισθών και των αμοιβών και σε περίπτωση που τέτοιοι κανόνες υφίστανται να επιβληθεί ή να είναι καλύτερη η επιβολή τους. Βεβαίως πολλά έχουν γίνει μέχρι τώρα για την ε, ισότητα όσον αφορά τις πολιτικές απασχόλησης. Όμως ακόμα βρισκόμαστε μακριά από το στόχο μας. Οι γυναίκες και οι άνδρες σαφέστατα δεν είναι ακόμα ίσοι ε, στην αγορά εργασίας και βεβαίως μεγαλύτερο τροχοπέδι ακόμα ε, σε αυτή την κατάσταση είναι η κρίση. Αυτά ήθελε να πει η Γκαμπριέλ Ζήμερ όσον αφορά την έκθεσή της. Βεβαίως αναμένω με τα σχόλιά σας. Δυστυχώς, δυστυχώς, ε, θα πρέπει να φύγω στη διάρκεια της συζήτησης, αλλά έχω συναδέλφους που θα παρακολουθήσουν και θα πάρουν ε, σημειώσεις. Ωραία, θα περιορίσουμε το χρόνο. Ένα λεπτό καθένας, παρακαλώ. Η κυρία Λόπεθ Φοντανιέχη τα κύρτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα μιλήσω πολύ γιατί πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε για αυτό το θέμα. Ότι οι γυναίκες πρέπει να πληρώνονται το ίδιο με τους άντρες για την ίδια δουλειά. Οι γυναίκες μπορεί καταρχήν επηρεάστηκαν λιγότερο από την κρίση, μάλλον γιατί είχαν χαμηλότερο επίπεδο θέσεις απασχόλησης από ότι άντρες. Τώρα όμως πλήττονται το ίδιο και ακόμα περισσότερο. Αλλά εγώ θέλω να μιλήσω εδώ κυρίως για τα προβλήματα των παιδιών, για την φτώχεια των ε, παιδιών. Γιατί οι γυναίκες που δεν έχουν ε, καλά αμοιβόμενη δουλειά ε, δεν μπορούν να προσφέρουν αρκετά και στα παιδιά τους. Η Ελισαβέτ Μωράν που είναι επί της ουσίας αρμόδια εισηγήτρια μιλάει για όλα αυτά, για τις γυναίκες και την απασχόληση. Οπότε η συγγήτρια βέβαια δύσκολα μπορεί να τα προσθέσει αυτά, μια που συμπεριλαμβάνονται. Οπότε πιστεύω ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε κάλλιστα το κείμενο αυτό και να συνεργαστούμε πλήρως με την κυρία Τσίμερ. Πρόεδρος, η κυρία Κλήφτη, πρώτα απ' όλα, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ. Όπως ξέρετε, είμαι σκιώδης συγγήτρια από πλευρά της Επιτροπής μας για αυτό το μεγάλο θέμα που με απασχολεί πολύ. Ούτε εγώ έχω πολλά πράγματα να προσθέσω, μόνο ότι έχω ετοιμάσει διάφορες τροπολογίε για το γυναικείο πρόσωπο της φτώχειας. Η συγγήτρια το λέει εδώ και καιρό. Δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα δυστυχώς, δεν έχουν γίνει βελτιώσεις. Ορισμένα φαινόμενα επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά. Μπορούμε κάλλιστα να τα αναλύσουμε εδώ. Να δούμε δηλαδή τη διάσταση άντρες, γυναίκες και όλες τις πολιτικές που έχουν να κάνουν με την απασχόληση. Πώς θα βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και την ευελιξία στην εργασία. Έπειτα να δούμε και την μακροοικονομική διάσταση σε σχέση με τον, την κοινωνική. Τι γίνεται στην αγορά εργασίας να μιλήσουμε ακόμα και για την πράσινη οικονομία που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά όταν ψάχνει μια γυναίκα δουλειά. Έπειτα ε, οι δημοσιονομικοί μηχανισμοί πρέπει να σέβονται τη διάσταση γυναίκα και να μην ξεχνάμε και τη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων, κυρίως όταν πρόκειται για αποφάσεις σε σχέση με την αγορά εργασίας. Κάποιες συνέπειες όμως δεν έχουν αναφερθεί σχεδόν καθόλου. Οι αλλαγές που γίνονται στις οικογένειες των εργαζόμενων αυτών γυναικών. Θα σας δώσω το παράδειγμα της δικιάς μου χώρας, της Ρουμανίας η ανεργία που πλήττει τις γυναίκες ε, δεν είναι τόσο ψηλή όσο εκείνη των ανδρών. Γιατί όμως, γιατί πολλές γυναίκες έφυγαν από τη χώρα και πήγαν να βρουν δουλειά αλλού στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό όμως δημιουργεί τεράστια προβλήματα για τα παιδιά τα οποία παραμένουν στη Ρουμανία και τα οποία τα φροντίζουν είτε συγγενείς είτε πάνε σε ιδρύματα. Ακόμα όμως και εκεί που γυναίκες δεν πλήττονται τόσο πολύ από την κρίση, και εκεί υπάρχουν οικογενειακές συνέπειες, σαν και αυτές που σας είπα. Γι' αυτό πρέπει να δούμε από κοντά το θέμα της ανεργίας για να υπάρχει καλύτερη ισορροπία, δηλαδή μεταξύ των εργού πληθυσμού να έχουμε εξίσου άντρες και γυναίκες. Σε τομείς όπως είναι οι υπηρεσίες όπου οι γυναίκες απασχολούνται εκεί περισσότερο, ε, προστατεύονται πιο πολύ από τις άλλες τομείς που παραδοσιακά είναι αντρικοί. Και μην ξεχνάμε και τις νέες γυναίκες, οι οποίες πρέπει να υποστηριχτούν για να μπορέσουν να βρουν δουλειά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ο Βίκε Μπαστός, η οποία εκπροσωπεί την κυρία ε, Μόρα Μπαστός. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κυρία Τζίμερ για την εργασία της, ε, για ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Σε γενική δεδομένη συμφωνώ με την ε, γνωμοδότηση της εισηγητρίας, η οποία αφορά την ισότητα των φύλων και διάφορα άλλα επιμέρους ε, ζητήματα. Δεν νομίζω ότι το κράτος θα πρέπει να τα ρυθμίζει όλα αυτά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δουλέψουμε σε βάθος Σήμερα το πρωί συζητήσαμε την έκθεση αυτή την, ε, στην Επιτροπή Γυναικών και ήταν ε, έτσι πολύ καλή η άποψη. Ρεζινά Μπαστός, εξ ονόματος της κυρίας Μωρές Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πραγματικά εξ ονόματος και συναδέλφου Ευρωβουλευτού θέλω να δώσω μια αξιολόγηση για την έκθεση της συναδέλφου Τσίμερ όπου από πλευρά ε, της ε, εισηγητρία Σάτιε από την Επιτροπή Γυναικών για την γνωμοδότηση για αυτή την έκθεση συμφωνεί με τι γενικέ γραμμές. Δεν έχει κάποια αντίθεση. Μάλλον συμμερίζεται κιόλας ε, την πρωτοβουλία για την πλατφόρμα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και συμμερίζεται την άποψη για την αδικία της συναδέλφου Τσίμερ, για τις δυσκολίες που υπάρχουν για τις γυναίκες για να έχουν πρόσβαση σε απασχόληση και εργασία ποιότητας, αναβαθμισμένες εργασίες ε, και τα κράτη-μέλη πρέπει να ενισχύσουν, να ε, ενδυναμώσουν την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση και να μπορέσουν οι περικοπές στις, στα δημόσια κονδύλια να ε, πάψουν ώστε να, υπάρξει, να μην επιδεινωθεί η κατάσταση της φτώχειας για τις γυναίκες. Από πλευρά τη κυρία ε, για την παρουσίαση αυτή που, είχα την που είχαμε την ευκαιρία παρουσίαση στην Επιτροπή Γυναικών, ε, φυστάται η προσοχή ότι σε αυτή την κρίση την οικονομική και χρηματοπιστωτική που δεν έχει κανένα παράλληλο ιστορικά από την εποχή του 1930, δεν θα πρέπει να εμβαθυνθούν οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτή η καταπολέμηση των ανισοτήτων σε σχέση με τα δύο φύλλα θα ε, πρέπει να αντιμετωπιστεί για να μην υπάρξει οπισθοδρόμηση και γίνεται αναφορά στο ότι άμεσα πλήττονται και οι άνδρες από αυτή την κατάσταση αλλά οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επίσης τα επίσημα στοιχεία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτό το στοιχείο γιατί οι γυναίκες όταν αποσύρονται από την αγορά εργασίας απασχολούνται με μη ανταμοιβόμενη εργασία ή προσωρινή εργασία επισφαλού, επισφαλούς χαρακτήρα. Επίσης ε, μια επισήμαση που γίνεται από πλευράς της κυρίας Σάτια για το θέμα της ε, αύξησης ουσιαστικά της ε, βίας εις βάρος των γυναικών σαν συνέπεια της κρίσης ε, που ζούμε. Ευχαριστώ. ο συνάδελφος που εκπροσωπούσε την κυρία Τζίμερ έχει φύγει. Εν πάση περιπτώσει, Υπάρχουν ε, οι πολιτικοί υπάλληλοι της ε, ομάδας ΓΚΟΕ που θα δώσουν όλα τα στοιχεία. Και, εν πάση τόσο, υπάρχουν δυνατότητες τροπολογίες που θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 8 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξετάσουμε τις ε, τροπολογίες αυτές που μπορούν να υποβληθούν μόνο στα αγγλικά. Παρακαλώ να το σημειώσετε αυτό, μόνο στα αγγλικά. Στις 14 Ιανουαρίου 23 Ιανουαρίου ενδεχομένω του συμβιβασμού, έτσι ώστε να ψηφιστούν 24 στην Επιτροπή. Η ΔΕ Επιτροπή Γυναικών ε, θα, πάρει την τελική της, ε, θα κάνει τελική ψηφοφορία 18-19 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, ε, δεν το συνηθίζουμε, αλλά παρόλα αυτά να σας πω ότι να θεωρήσουμε τροπολογίες 11, μάλλον τα σημεία ενώ η Πρόεδρος, 11 και 12 είναι σημεία ε, προς πληροφόρηση ε, και η διαδικασία πληροφόρησης θα γίνει γραπτά. Επομένως, και όσον αφορά τη διαπραγματεύση με το Συμβούλιο σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και όσον αφορά τις ε, ε, διαπραγματεύσεις, συγγνώμη, την αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αποσχόλησης ε, στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας στη Γενέβη στις 12 Ιανουαρίου του 2012. Αυτές οι πληροφορίες θα σας δοθούν γραπτά. Σημείο 7 λοιπόν της ημερησίας διατάξεως. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον Στίφεν Χιούζ, ο οποίος είναι εισηγητής για έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με απειλές κατά της υγείας στο χώρο εργασία λόγω αμοιάντου και προοπτικέ εξάλληψη του αμοιάντου που εξακολουθεί να υφίσταται. Πρόκειται για 120 τροπολογίες οι οποίες έχουν υποβληθεί στην έκθεση αυτή. Κύριε Ισηγητά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές. Ε, καμιά φορά το κάνουμε έτσι λίγο τυπικά. Εγώ το εννοώ, τους ευχαριστώ όλους τους σκιώδεις εισηγητές ε, για, αυτές ε, τις, ε, για τις προτάσεις που κάνανε, για τις τροπολογίες τους, ε, στις συναντήσεις που είχαμε. Τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ καλά, η συνεργασία ήταν εξαιρετική. Θα κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις στην αρχή. Πρώτα απ' όλα ότι εδώ πρόκειται για μη μαθητικό κείμενο, δηλαδή είναι μια πρόταση πρωτοβουλίας Εμεί Εμείς προσπαθήσαμε σε ένα-δυο σημεία να προωθήσουμε τα πράγματα, να τα σπρώξουμε πάρα πολύ. Γι' αυτό λοιπόν ε, ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να σπρώξουμε την Επιτροπή να κάνει μερικά βήματα προς εμάς και προς τη θέση μας. Όπως ε, είπατε κυρία Πρόεδρε υπάρχουν 120 τροπολογίες, περισσότερες εκ των οποίων με βρίσκουν σύμφωνο. Υπάρχουν τρεις ε, ε η κυρία Σέα και την κυρία Μακιντάιερ που δυσκολεύομαι να τις παρακολουθήσω. Ζητούν πολλές διαγραφές και για προφανείς λόγους βεβαίως δεν μου αρέσουν οι τροπολογίες τους. Είμαι, σχεδόν, είμαι κατά σχεδόν όλων των τροπολογιών τους. Επίσης έχω κάποιες δυσκολίες με τις τροπολογίες του Ρόζα Χέλμερ. Διότι εκείνος προσπαθεί να ε, να υποβαθμίσει τα προβλήματα υγείας τα οποία προκύπτουν από τη χρήση λευκού αμοιάντου. Ε, και νομίζω ότι αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Είναι ε, εξίσου ε, σημαντικά τα προβλήματα με αυτά που προκαλούν και ο καφέ και ο κιανούς αμίαντος και επομένως δεν μπορώ να δεχτώ αυτά τα, αυτές τις τροπολογίες. Πέραν των τροπολογιών που έχουν υποβληθεί από αυτούς τους τρεις συγητές, μπορώ να συμφωνήσω μάλλον με τους περισσότερους από τους υπολείπους ε, συμφωνήσαμε όλοι ότι ο αμίαντος είναι σημαντικό πρόβλημα υγείας, ε, επίσης ότι θα πρέπει ε, να, πρέπει, θα πρέπει να αναγνωριστούν καλύτερα και ομοιόμορφα οι ασθένειες οι οποίες οφείλονται στην έκθεση σε αμίαντο, επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες κοινέ διατάξεις όσον αφορά τη διάγνωση. Υπάρχουν 15 κοινέ τροπολογίες από τον George Μπακ, τον υποφαινόμενο, ε, την συνάδελφο Μωρίνη Σαντιέν και ε, τον συνάδελφο Και ενσωματώνονται βεβαίω στην έκθεση. Επίσης ε, έχουν προετοιμαστεί, έχω προετοιμάσει μάλλον 15 συμβιβαστικές τροπολογίες οι οποίες περιλαμβάνουν την μεγάλη πλειοψηφία των υπολείπων υποβληθισών τροπολογιών. Έχουμε τέσσερις ομάδες ε, οι οποίες έχουν ε, ασχοληθεί με τις ε, τροπολογίες αυτές. και λάβαμε κάποια, ένα, κάποια mail σήμερα το πρωί από τον σκιώδη των φιλελευθέρων που προτείνει κάποιες αλλαγές σε πέντε από τις συμβαστικές τροπολογίες. Νομίζω ότι στις δύο υπάρχει ήδη συμφωνία. Περιμένω και την άποψη των άλλων σκιωδών για να δούμε αν ε, μπορούμε να δεχτούμε ε, τις τροποποιήσεις αυτές όσον αφορά τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Δεν έχω ακόμα το απαραίτητο feedback από τους υπολείπους. Έχουμε λοιπόν συμφωνία όσον αφορά τους άλλους, Ανδρέα Ζαμόνη και ο... With, um, all, if not all, then practically all of the amendments that they have suggested. So I think um, we have a, a large degree... Ε, γενικώς για τους άλλους ε, νομίζω ότι μπορούμε... Ε, ναι, είδε και οι τροπολογίε του κυρίου Πουπάκη που επίση θα πρέπει να ζητηθούν λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε. Τον Στίβεν Χιούς, τον συνάδελφο, για αυτή τη φιλόδοξη έκθεση πρωτοβουλίας να τον ευχαριστήσω. Και όσον αφορά τη συνεργασία μπορώ να ανταποδώσω τον έπαινο, τους επένους. Ευθύ εξ αρχή υπήρχε καλή ενημέρωση σε τακτά διαστήματα και στι δύο συναντήσει που είχαμε συζητήσαμε ανοιχτά και ειλικρινά και προ όφελο ε, τη έκθεση. Και έτσι έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα τελικά. Από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Πιστεύω ότι ευθυγραμμίζεται και με τη δική μας γνωμοδότηση αυτή η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Σε κάποια σημαντικά σημεία θέλω να επικεντρωθώ και να τα τονίσω. Το θέμα του screening, της εξέτασης ε, και της ε, καταχώρησης. Ε, καλοί συμβιβασμοί βρέθηκαν. Το ΕΛΚ υποστηρίζει επίσης την πρόταση Steven Hughes για τον καθορισμό μιας ημερομηνία. Μέχρι πότε δηλαδή τα δημόσια κτίρια θα πρέπει από τα δημόσια κτίρια να αφαιρεθεί ο αμίαντος. Και υποστηρίζουμε επίσης και τη σύσταση για τη δημιουργία δημόσιων μητρών ή καταλόγων ε, για τον ε, ε, αμίαντο από τα κράτη-μέλη. Στην παράγραφο 12 για την ανάπτυξη προγραμμάτων εξυγίανσης κάποιες μικρές λεπτομέρειες πρέπει να αποσαφινιστούν, αλλά πιστεύω ότι και εκεί μπορούμε πάλι να συμφωνήσουμε τελικά. Είναι, ας το πω έτσι, κάποιες ερμηνείες επί του κειμένου που προκαλούνται από, τη μετάφραση κάποιων παραγράφων. Μια σημαντική συμφωνία βρέθηκε στη διασφάλιση των προσόντων και της κατάρτισης παράγραφοι 9 και 10 που απαιτούν στο μέλλον ελάχιστες προδιαγραφές να ισχύουν για συγκεκριμένα προσόντα και ε, ε, ε, ικανότητες όσον αφορά τον αμίαντο και με ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τους εργαζόμενους που εργάζονται σε περιβάλλον αμοιάντου. Νομίζω είναι καλές οι προϋποθέσεις για αυτή την έκθεση να μην ενδυναμωθούν οι προτάσει αυτές μέσω των διαπραγματεύσεων. Είναι φιλόδοξο αυτό το εγχείρημα και έτσι αυτό πρέπει να γίνει από πλευρά να ευδοκιμήσει η έκθεση πρωτοβουλία. Βρίσκει ευρύτερη υποστήριξη και σίγουρα όσον αφορά τι ε, παρεμβάσει που χωρίς εξαίρεση προς αυτή την κατεύθυνση πορευόμαστε. Πριν από τις διακοπές ή αμέσως μετά από τις διακοπές θα αναφέρουμε τα σχετικά για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ και πάλι και σίγουρα θα είναι μια πολύ καλή έκθεση. Ευχαριστώ. Ε, Κάρι Μαντελή και μετά κύριο Σκάρκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα στον εισηγητή μας πρώτα απ' όλα που ζήτησε τη συμμετοχή μας σε όλες τις ε, συνεδριάσεις προκειμένου να ετοιμαστούν οι συμβαστικές τροπολογίες. Εμείς οι οικολόγοι συμφωνούμε με όλες τις τροπολογίες που υποβάλλει. Βέβαια ακόμα δεν είχα την ευκαιρία να κοιτάξω αυτά που υπέβαλε ο κύριος Πινιόν. Αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι τον εισηγητή για τις τροπολογίες. Την τροπολογία, ο, θέλει να την ε, διαγράψουμε. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν κρίμα. Θα μπορούσατε να μου απαντήσετε σε αυτό παρακαλώ. Παράγραφος 17, δηλαδή τροπολογία ο, ο. και μετά Φιλμπενιάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλάμε για τον αμύαντο. Βέβαια, όλες οι ουσίες έχουν διαφορετικές μορφές. Υπάρχει ο μπλε, ο καφέ και άσπρος. Οι πρώτοι έχουν ε, θανατηφόρες επιπτώσεις μακροπρόθεσμα στους πνεύμονες που τους καλύπτουν και γι' αυτό και στο τέλος είναι θανατηφόρα η ενώ ο λευκός έχει να κάνει με τον μαγνήσιο, είναι κάτι εντελώ διαφορετικό. Και δεν βλάπτει την υγεία. Και δεν επηρεάζει μακροπρόθεσμα αυτούς οι οποίοι αναπνέουν τα σωματίδια αυτού του είδους του αμίαντου. Το 1997 σε έκθεση ο καθηγητής Πέτο κάνει ένα στατιστικό σφάλμα γιατί λέει ότι 90% του αμοιάντου που χρησιμοποιείται είναι λευκός. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Είναι λάθος. Και αργότερα η υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου για την ασφάλεια και την υγιεινή όσον αφορά την τοξικολογία λέει ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία από τον ε, αμίαντο που χρησιμοποιείται στο τσιμέντο. Από τον λευκό λοιπόν αμίαντο δεν υπάρχουν κίνδυνοι, ενώ από τον μπλε και τον καφέ ναι. Παρόλο λοιπόν που θέλουμε να αποδαιμονοποιήσουμε τον ε, λευκό αμίαντο, παρόλα αυτά υπάρχει μεγάλο λόμπι υπό τη Λόρη Καντζάνα Λάρν για παράδειγμα στον Ηνωμένο Βασίλειο που είναι αδερφή του επικεφαλής ενός ε, εταίρου σε μια εταιρεία στην ε, Καλιφόρνια που κερδίζει εκατομμύρια και εκατομμύρια από το εμπόριο αμίαντου. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τον λευκό αμίαντο. Ε, ο κρυσταλλώδης ξαλώδες μαγνήσιο είναι αυλαβές και συμπεριλαμβάνεται ε, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα σε διάφορα μείγματα, σε αντίθεση με το μπλε και το καφέ. Αν εμείς αποφασίσουμε να εξαφανιστεί πλήρως ο αμύαντος, τότε οι επιπτώσεις είναι τεράστιες. Γιατί έχετε πάρα πολλούς που θα επηρεαστούν από μια τέτοια απόφαση, από δικηγόρους, γιατρούς, ε, εργαζόμενους. Το κόστος της αφαίρεσης του αμοιάντου, παντός είδους αμοιάντου από παντού, θα έχει τεράστιες επιπτώσεις και θα κοστίσει πάρα πολλά χρήματα. Θα επηρεάσει πάρα πολύ την ευρωπαϊκή οικονομία. Οι αγρότες δε θα επηρεαστούν πάρα πολύ γιατί έχουν πάρα πολλά κτίσματα με αμίαντο. Αν λοιπόν περάσει η έκθεση αυτή, μπορείτε να περιμένετε να δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα και να έχετε εναντίον σας όλο το λόμπι των ε, γεωργών. Ολοκληρώστε παρακαλώ, διακόπτη πρόεδρος. Ναι, θα υπάρξει και επιπλέον κόστος, γιατί να αφαιρέσετε τον αμίαντο, θα πρέπει να απαλλαγείτε από αυτόν. Σε χωματερές, και πρέπει να τον αντικαταστήσετε βέβαια με άλλα πιο σύγχρονα υλικά, τα οποία δεν τα ξέρουμε ακόμα. Δεν πρέπει να περάσει η έκθεση αυτή έτσι ως έχει κυρία Πρόεδρε. Φίλ Μπινιό που είναι ο τελευταίος μιλητής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή για τον ε, επικοδομητικό διάλογο που είχαμε μεταξύ μας. Μπορέσαμε έτσι να επεξεργαστούμε πάρα πολλά θέματα και τώρα αντιλαμβάνομαι ότι μιλάμε μόνο για τα δημόσια κτίρια. Αυτή είναι η πρότασή του. Και αυτό ακριβώς γιατί υπήρξαν τροπολογίες για να εξαιρεθούν τα γεωργικά κτίσματα που συμπεριλαμβάνονταν στην αρχή. Το αλλάξαμε αυτό. Υπάρχει λοιπόν ένας συμβιβασμός που το λύνει αυτό το ζήτημα. Διαβάστε το καλύτερα κύριε συνάδελφε και όλοι οι υπόλοιποι πριν ψηφίσουμε για να βεβαιωθείτε για αυτό που σας λέω. Ο κύριος Γιούς αναφέρεται στις αλλαγές που ζητάω και εγώ με τους συμβασμούς. Μερικές αλλαγές δεν έχουν μεγάλες επιπτώσεις. Πρόκειται για μια λάθος λέξη που χρησιμοποιείται για παράδειγμα. Η συμβαστική ΚΚ δεν νομίζω ότι είναι τόσο επίμαχη. Πρόκειται για το άρθρο 14 της προηγούμενης οδηγίας. Το άρθρο αυτό λοιπόν μιλάει για την προηγούμενη οδηγία και εμείς θέλουμε να διευκρινίσουμε περί τίνου σε πρόκειτο ακριβώς. Για τη συμβαστική L επίσης, και εδώ προτείνουμε κάποιες αλλαγές. Η πρώτη είναι να αφαιρεθεί το manages. γιατί καλύπτεται από τις οικοδομικές δραστηριότητες αναφερόμασταν τότε στη διαχείριση του αμοιάντου. Το management πήγαινε στον αμοιάντο και όχι στις επιχειρήσεις, οπότε υπήρξε μια λάθος ερμηνεία όσον αφορά την αρχική τροπολογία, γι' αυτό και το αλλάξαμε εκεί. Έπειτα προτιμάμε το as appropriate στην κατάρτιση, γιατί δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνει κανείς την κατάρτιση αν είναι ενός είδου και δεν χρειάζεται παραπέρα. το L και στο M. Το αφήνω λοιπόν στον εισηγητή να μας πει ποια είναι η γνώμη του. Εμείς προτείνουμε να βάλουμε should. Θα έπρεπε. Γιατί και εδώ υπάρχουν πολλές, ε, υπάρχουν μάλλον οι χώρες μέλη που έχουν αρμοδιότητα. Η μεγαλύτερη πάντως διαφορά μας έγινε στην τροπολογία G. που μιλάει για την ημερομηνία 2028. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτή την ημερομηνία. Γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο λογαριασμός που θα πρέπει να πληρώσουμε, πόσο θα κοστίσει. Σε πολλές χώρες μέλη θα διαπιστώσουμε ότι έχουν πάρα πολλά κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία και άλλα δημόσια κτίρια που χτίστηκαν τη δεκαετία του 60 και του 70 τότε που χρησιμοποιόταν πάρα πολύ αμύαντος. Δεν έχουμε ιδέα δηλαδή τι προτείνουμε τελικά αν βάλουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία προκειμένου να έχει αφαιρεθεί μέχρι τότε ο αμύαντος. Προτείνουμε λοιπόν να γίνει πρώτα μια έκθεση αντικτύπου, να δούμε ποιο θα είναι το κόστος και το όφελος και μετά να αποφασίσουμε. Εξαλλού αυτή την πληροφορία μπορούμε να την έχουμε γρήγορα. Αν θέλουμε να ξέρουμε πόσα σχολεία, πόσα νοσοκομεία, πόσα θα μας κοστίσει, στις διάφορες χώρες, θα θέλουμε κάπου δύο χρόνια για να πάρουμε την πληροφορία αυτή. Οπότε να ξέρουμε τι ζητάμε. Μην βάλουμε ημερομηνία, αν προηγουμένως δεν ξέρουμε πόσο θα μας κοστίσει. Αυτό που θα προτιμούσα εγώ είναι μια πραγματιστική, έτσι, ρεαλιστική προσέγγιση όσον αφορά την αφαίρεση του αμοιάντου. Βλέπετε, πολλά από τα κτίρια αυτά, έτσι αλλιώς είναι κτίρια, τα οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να καταδεφιστούν. Οπότε προτιμάμε σε αυτή την περίπτωση να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που θα γίνει είναι ότι όταν φτάσουν σε σημείο κατεδάφιση τα κτίρια αυτά, τότε να έχουμε την εγγύηση ότι ο αμίαντος θα αφαιρεθεί και θα απομακρυνθεί με ασφάλεια για την υγεία των ε, πολιτών. Και μην ξεχνάτε ότι παίρνουμε πολλές και διάφορες αντιφατικές πληροφορίες και ολοκληρώνω με το τελευταίο μου. Παίρνουμε λοιπόν εντελώς διαφορετικές πληροφορίες, προς διαφορετική κατεύθυνση όσον αφορά τον αμίαντο. Έχουμε επιστήμονες που λένε το ένα και άλλους επιστήμονες που λένε το άλλο. Οπότε, α ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ, να μας το διευκρινίσει αυτό ή, εν πάση περιπτώσει, να κάνει κάποια δουλειά για να καταλήξει σε μια αξιόπιστη μελέτη και μια αξιόπιστη απάντηση. Προς το παρόν σας είπα, έχουμε αντιφατικές πληροφορίες και δεν μπορούμε να αποφασίσουμε κάτω από αυτούς τους όρους. Πρόεδρος, θα κλείσω τον κατάλογο των... Ε, τον έκλεισα μάλλον των ομιλητών. Να απαντήσει ο συγητή παρακαλώ λίγο γρήγορα γιατί περνάει ο χρόνος, δεν προλαβαίνουμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδες για τα σχόλια που έκαναν ε, να ασχοληθώ με ένα-δυο σημαντικά θέματα όσον αφορά τον ε, λευκό αμμίαντο, το, το, δηλαδή. Εμείς έχουμε την άποψη ότι και οι τρεις μορφές του αμιάντου αυτή τη στιγμή που βρίσκονται εκτός νομοθεσίας, νομοθετικού πλαισίου ε, ε, και είναι παράνομοι και οι τρεις μορφές για την Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένως ε, θα πρέπει να έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Και εγώ μπορώ να σας παρατάξω μια σειρά εκθέσεων και έρευνων που έχουν άλλου είδους αποφάσεις. Ε, στην Ιταλία, ας πούμε, ε, έχουμε ε, έρευνα η οποία καταδεικνύει ότι υπάρχουν 27 θάνατοι από χρήση, ίνες, από χρήση ινών χρυσοτελικού αμοιάντου. Επομένως, είναι εξαιρετικά επικίνδυνος ο αμίαντος αυτός. Λαμβάνουμε υπόψη μας... Ε, λαμβάνονται υπόψη ε, βεβαίω ε, και μελέτες που έγιναν στο ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο και δημοσιοποιήθηκαν πριν από 7 χρόνια όπου αναφέρονται και ο Κιανού και ο, καφέ και ο λευκός Αμίαντο ως έχοντες την ίδια επικινδυνότητα. Κοιτάξτε, εάν δεν είναι σαφή τα πράγματα, νομίζω ότι μέσω των ε, συμβιβαστικών τροπολογιών μπορούμε να τα κάνουμε σαφε, σαφέστερα. Ε, όσον αφορά τις, ε, τους συμβασμούς I και K, θα συζητήσω λοιπόν με τους σκιώδεις. Όσον αφορά το G, ε, του προτείνω να το ξαναδούμε, να καθίσουμε να το ξαναδούμε, γιατί βεβαίως οποιαδήποτε ε, πρόταση η οποία αφορά ε, την Κομισιόν φυσικά θα υποβληθεί σε μελέτη αντικτύπου. Τώρα, αν πρέπει να το αναφέρουμε ρητά, δεν είμαι και βέβαιος, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να δω και τι feedback θα μου δώσουν οι σκιώδεις εισηγητέ. Αυτά, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, κυρία Πρόεδρε, ξέρω ότι δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, αγαπητέ συνάδελφε. Επομένως, ολοκληρώσαμε και με τον έλεγχο των τροπολογιών επί της εκθέσεώς σας. 24 Ιανουαρίου θα εγκρίνουμε τη γνωμοδότηση για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε το Φεβράριο στην Ολομέλεια. Ίσως θα πρέπει να μας αποσαφηνίσει και η Κομισιόν εκτός όμως ε, της ε, αιθούσης σχετικά με τις απόψεις της όσον αφορά το λευκό αμίαντο σημείο 8 της ημερησίας διατάξεως και θα δώσω αμέσως το λόγο στην Βερόνικα Λόπε Φοντανιέ για να μας μιλήσει για τις 256 τροπολογίες που έχουν υποβληθεί ε, για την έκθεσή της για το εξάμεινο συντονισμού. Δεν θα μας τις ε, παρουσιάσετε φαντάζομαι όλες, ε, θα δείξετε συνθετικό πνεύμα. Ευχαριστώ πολύ και βεβαίως ε, πρέπει να μελετηθούν με μεγαλύτερη ηρεμία. Αυτό θα κάνω κατά τη διάρκεια των διακοπών του, των Χριστουγέννων, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιτύχουμε συνολική συμφωνία. Θα συνεχίσω στα Ισπανικά τώρα. Θέλω να πω λοιπόν ότι προσπαθώ με το κείμενό μου, με τη βοήθεια όλων, να συμπεριλάβω όσο γίνεται περισσότερες από τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν στις συμβαστικές μου τροπολογίες. Και είναι πολύ σημαντικό, το έχω ξαναπεί, η έκθεση αυτή δεν, με την έκθεση αυτή δεν φαίνεται ξεκάθαρα ποιος έχει την αρμοδιότητα. Πάντως αν εμείς εγκρίνουμε με μεγάλη πλειοψηφία την έκθεση αυτή, τότε η νομιμότητά μας ενισχύεται για αυτό το θέμα. Γι' αυτό να την κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια και εγώ βέβαια πρώτη από όλους. Προσπαθούμε να είμαστε ευέλικτοι ώστε όλες οι πολιτικές ομάδες να συμφωνήσουν τελικά. Με τις συμβαστικές τροπολογίες αυτό ακριβώς προσπαθούμε να πετύχουμε. Η έκθεση είναι λίγο μεγάλη, Χρέστηκε να προσθέσω διάφορα, αλλά δεν θέλω να προσθέσω ακόμα πιο πολλά με τις συμβαστικές τροπολογίες. Ίσως να αφαιρέσω και να αντικαταστήσω κάποια κομμάτια της έκθεσης από τις συμβαστικές τροπολογίες για να μην βαρύνει υπερβολικά, να μην είναι υπερβολικά μεγάλη. Να συνεχίσει να υπάρχει συνοχή πάντως. Θέλω ακόμα να διευκρινίσω ότι εδώ πέρα τίθεται θέμα και πολιτικών προσανατολισμών, χωρίς βέβαια να βάζουμε λεπτομέρειες. Υπάρχουν τροπολογίες που είναι πολύ πλήρεις και θα μπορούσαν από μόνες τους να αποτελέσουν αντικείμενο έκθεσης πρωτοβουλίας. Για παράδειγμα, εκείνες οι οποίες αναφέρονται ε, στους νέους. Αλλά, όπως είπα και πριν, πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε την έκταση του κειμένου μας και να περιοριστούμε στους γενικούς προσανατολισμούς. Έτσι καλώς θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στη συνεδρίαση των ε, σχεδόν εισηγητών. Τώρα έρχομαι πάλι στις συμβαστικές τροπολογίες. Σε κάποιες τροπολογίες λέμε ότι πρέπει να υπογραμμιστεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων και να ενισχυθεί μάλιστα ο ρόλος τους. Αυτό μπορούμε να το συμπεριλάβουμε. Επίσης, όταν μιλάμε για την απασχόληση και την ευελιξία στην εργασία, λένε κάποιες τροπολογίες ότι πρέπει να τονίσουμε περισσότερο την σταθερότητα. Ναι, μεν ελαστικότητα, αλλά και σταθερότητα στην ε, απασχόληση. Και αυτό πρέπει λοιπόν να το συμπεριλάβουμε στις συμβαστικές τροπολογίες. Όσο αφορά τώρα το φορολογικό, σίγουρα έχει επιπτώσει στη δημιουργία ή στη μη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Χρειάζεται λοιπόν φορολογική σταθερότητα και Γι' αυτό οι τροπολογίε οι οποίε δεν το θέλουν δεν με βρίσκουν σύμφωνοι. Πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στη λιτότητα και στην ανάπτυξη κάποια ισορροπία. Πάντως πιστεύω ότι θα καταφέρουμε μεταξύ μα όλοι να καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική για όλους διατύπωση. Μεταξύ άλλων γιατί η κατάσταση στι χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαφορετική ε, από χώρα σε χώρα και άρα πρέπει να προσαρμόζεται κάθε χώρα ανάλογα με την κατάσταση της απασχόλησης ή της ανεργίας εκεί. Τέλος, να ευχηθώ καλές γιορτές σε όλους. 7 Ιανουαρίου ραντεβού με τους σκιώδεις συζητητές, εκείνη τη βδομάδα δηλαδή. Έχουμε πολλή δουλειά και λίγο χρόνο. Ας επωφεληθούμε λοιπόν για να διαπραγματευτούμε πάνω στις συμβαστικές αυτές τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρόεδρος, θα περιορίσω το χρόνο ομιλίας τώρα. 1,5 λεπτό καθένας. Κουτιέρες ε, Πιώτο και μετά Χάρκιν. Ή ε, μάλλον... Α, πήγε να αρχίσει η κυρία Χάρκιν. Όχι, λάθος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Ο ο στόχος μας πρέπει να είναι σαφής με την έκθεση αυτή. Πρέπει να είμαστε άκαμπτοι όσον αφορά την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια διαφορετική οικονομική πολιτική που τη ζητάμε. Είπε η συγκήτρια ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφιβολίες για τις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας, για την ε, στάση μας. Ναι, αλλά ολόκληρη η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επηρεάζει την απασχόληση και την ποιότητα της απασχόλησης. Για τους σοσιαλιστές υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές που θέλουμε να τις ξεκαθαρίσουμε ευθύ αμέσω. Το ένα έχει να κάνει με την ελαστικότητα. Κοιτάξτε, σε πολλές χώρες, εκεί που υπάρχουν ε, τέτοια μέτρα, πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο δημοσιονομικός φάκελος ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί τελικά και να είναι σύμφωνος με το σύμφωνο σταθερότητας. Μετά το τελευταίο συμβούλιο φαίνεται γιατί για τον χρυσό κανόνα του να μην ληφθούν υπόψη τομείς όπως είναι η απασχόληση, η εκπαίδευση, να μην λαφθούν οι υπόψη τους όταν γίνονται δαπάνες παρά το έλλειμμα που μπορεί να έχουν οι προπολογισμοί των χωρών και να φροντίσουμε για τη δημοκρατική νομιμότητα όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στις μεταρρυθμίσεις των χωρών ε, μελών που πολλές φορές δεν είναι με διαφάνεια η Μαριάννα Χάρκιν. Και μετά Κορνέλισεν. Θα είμαι σύντομη. Πρώτα απ' όλα να πω στον εισηγητή ότι έχουμε εξαιρετικό έγγραφο εδώ, στην εισηγήτρια μάλλον, Πιστεύω ότι κάποιες από τι τροπολογίε ε, που, θα αναφέρω δεν είναι απαραίτητα δικές μου, πάντως στο θέμα ε, των λαμφα, λανθασμένων προβλέψεων και ο αντίκτυπο όπου αυτές μπορεί να έχουν θα πρέπει να συζητηθεί. Επίσης η δουλειά όσον αφορά την Προεδρία Κοινωνική, Διακυβέρνηση, Social Label ε, οι τροπολογίες ε, σημαντικές ε, άλλων και τις υποφάνημες Επίσης, όσον αφορά την δημοσιονομική εξυγίανση, αυτή θα πρέπει να είναι διαφοροποιημένη, θα πρέπει να είναι σωστή και θα πρέπει να είναι τέτοια που να μην καταστρέψει ακόμα περισσότερο την ίδια την σύνθεση, την κοινωνική της κοινωνίας μας. Νομίζω ότι όλα αυτά τα θέματα συνδέονται μεταξύ τους ε, και βεβαίως ε, η σύνδεση της παρούσας πολιτικής με την ετήσια, ε, την ετήσια έκθεση απασχόλησης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τελικό, τέλος, έκθεση προόδου του 2000, για το 2020 θα πρέπει οπωσδήποτε να ενσωματωθεί σε αυτό το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο Συνεργασμού των Οικονομικών Πολιτικών. Ευχαριστώ πολύ, ναι. Συμφωνώ απόλυτα με την προλαλήσαντα και αυτά. Θα ήθελα μόνο να αναφέρω την τροπολογία 48 να επιστήσω την προσοχή σας που στην αρχή, στην αρχή της έκθεσης ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προβούν σε μια διοργανική συμφωνία μαζί μας ως Ευρωβουλή ώστε να μας δώσουν ένα αξιόλογο ρόλο όσον αφορά αυτή τη διαργασία και με μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσαμε να έχουμε έναν ε, σπουδαίο ρόλο χωρίς να απαιτείται μια αλλαγή συνθήκης και να έχει νόημα αυτό το εγχείρημα. Αυτό πρέπει να είναι κλειδί για μας ε, για να πετύχουμε αυτή τη δυνατότητα. Όλα τα άλλα θα αποκτήσουν πρόσθετη αξία αν θα μπορούσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων. Ευχαριστώ. Ε, και εγώ χαιρετίζω την καλή και ισορροπημένη έκθεση με στοχοθέτηση ορθή από πλευράς εισηγήσεως και τις δυσκολίες που είχε λόγω της πιεστικής προθεσμίας. Το ίδιο ισχύει και για μας τους Ευρωβουλευτές. Με αυτή τη σημαντική έκθεση θα έπρεπε να μπορούσαμε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να συζητήσουμε. Ένα σημαντικό σημείο της εξυγίασης και παγίωσης των δημοσιονομικών στα κράτη-μέλη, καθένας είναι πεισμένος ότι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, αλλά θα έλεγα ότι και επανειλημμένα αναφέρθηκε πρέπει να μεριμνήσουμε για την ανάπτυξη. Ανάπτυξη. Διαφορετικά τεράστια κοινωνικά και δημοκρατικά προβλήματα θα αντιμετωπίσουμε μέσα στα, από πλευρά των κρατών μελών. Είναι παράδοση πλέον εν τω μεταξύ σε αυτή την έκθεση για την ανάπτυξη η κοινωνική πολιτική να έχει μια, ένα ρόλο στο περιθώριο. Πολλά αναφέρονται για τα δημοσιονομικά, τα οικονομικά, αλλά για τα κοινωνικά όχι. Πρέπει στις αντίστοιχες παραγράφους να αποφύγουμε την ε, ε, κοινωνική αποδόμηση. Και στην παράγραφο 33 για παράδειγμα εξεπλάγει για την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συντάσσει και λέει ότι ή δυνατόν η διασύνδεση του προσδόκιμου λέει ζωής και της ευημερία θα πρέπει να λειτουργεί με, κάποια, με κάποιο αυτοματισμό ώστε να αποφύγουμε λέει ε, αντιφάσεις σε ε, αντίθεση με τον παραδοσιακό κοινωνικό διάλογο όπου οι διαπραγματεύσεις για αυτά τα θέματα έχουν τεράστια σημασία. Ευχαριστώ. Euh, θα ξαναδώσω το λόγο στην εισηγήτρια, αλλά έχω κάτι που με απασχολεί. Δηλαδή ότι στη δική μας διαδικασία η γνωμοδότηση της Επιτροπής θα πρέπει να δοθεί με τις βέλτιστες συνθήκες και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει και η Επιτροπή νομικό, συγγνώμη, ε, Οικονομικών έτσι ώστε ε, να συνδυαστούμε όσο γίνεται περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Απλά και μόνο να ευχαριστήσω όσους παρανέβησαν. Πιστεύω ότι μια πολύ καλή δουλειά μπορούμε να κάνουμε και δεν θα μακρηγορήσω περισσότερο διότι θα πρέπει να συγκεκριμενοποιήσουμε τους συμβιβασμούς. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Merci. Euh, sur cette base, nous... Πολύ ωραία. Θα ψηφίσουμε λοιπόν στην έκτακτη συνεδρίασή μας στο Στρασβούργο στις 14 ε, Ιανουαρίου και θα φτάσουμε στην Ομέλεια 4 ε, με 7 ε, Φεβρουαρίου, ενώ εντωμεταξύ θα έχουμε και την Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Ομάδα. Ζητώ συγγνώμη από τους φιλοξενούμενους, αλλά πρέπει, είμαι υποχρεωμένη να εξετάσω ακόμα ένα ζήτημα πριν ξεκινήσουμε την ακρόαση. Στο σημείο 10 λοιπόν θα δώσω το λόγο αμέσως στη Γιούτα Στάινρουκ για να μας παρουσιάσει την γνωμοδότηση της Επιτροπής μας, της Επιτροπής ε, δηλαδή Απασχόλησης, ε, αυτή την ε, γνωμοδότηση που θέλει να υποβάλει στην Γιούρη όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2004-25 κάθετος Ευρωπαϊκή Κοινότητα σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς. Παρακαλώ, παρουσιάστε την γνωμοδότησή σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Σήμερα το πρωί η Νομική Επιτροπή συζήτησε για το θέμα του takeover bids. Και φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει η άποψη από πλευράς αυτής της Επιτροπής ότι η υφιστάμενη οδηγία δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί. Από την, τα κοινωνικά θέματα και τα θέματα της απασχόλησης βλέπω την ανάγκη τα δικαιώματα των εργαζομένων και η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων πρέπει να διασφαλιστεί και να εμπλουτιστεί περαιτέρω θα πρέπει οι γυναίκες και άνδρες εργαζόμενοι με συγχωνεύσεις ή αγορές να προστατεύονται καλύτερα, να έχουν ευρύτερα δικαιώματα, άμεση ενημέρωση, άμεση ενημέρωση και πληροφόρηση προς τους εργαζόμενους σε τέτοιες περιπτώσεις συγχωνεύσεων και το δικαίωμα στην απόφαση των κοινωνικών εταίρων να λαμβάνεται υπόψη πριν από τέτοιες αγορές ή συγχωνεύσεις. Αντίστοιχα, τη γνωμοδότησή μου έτσι τη συνέταξα λοιπόν, με αυτές τις κατευθύνσεις. Και στην περίπτωση που η οδηγία αυτή στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων επεξεργαστεί, ε, ε, εξεταστεί εκεί, θα έλεγα υπό το πρίσμα των πολιτικών για την απασχόληση θα πρέπει να ενταχθούν κάποιες πτυχές, ε, κάποια εδάφια σε αυτήν. Ολοκλήρωσα. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ζητά κανείς το λόγο, όχι, Ενάμιση λεπτό. Έχετε το λόγο. <clears throat> Um, Ευχαριστώ πολύ. Χρειάζεται ένα δίχτυ ασφαλεία όσον αφορά αυτέ τι προσφορέ εξ Αλλά θα πρέπει να στείλουμε κάποια σημάδια και λογικής αλλά και ε, σεβασμού των νομοθεσιών ε, στις χώρες ε, μέλη. Δεν περιμένουμε βέβαια ότι θα αλλάξουμε το νομοθετικό πλαίσιο των εξαγορών. Μπορεί να υπάρξει βέτο από τους κοινωνικούς εταίρους. Άρθρα 9, 10 και 12 μας δημιουργούν προβλήματα, εμένα τουλάχιστον προσωπικά. εμπλοκή και παρουσία των εκπροσώπων των εργαζομένων σε όλα τα στοιχεία. Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορεί όμως να μπλοκάρει την ε, εξαγορά απλά γιατί δεν τη θέλουν οι κοινωνικοί εταίροι. Το κόστος το οποίο ε, θα πρέπει να ενσωματώσει ε, των εκπροσώπων δηλαδή και των συνδικαλιστικών οργάνων που θα πρέπει να ενσωματωθεί. Δεν καταλαβαίνω γιατί μπορώ να, πρέπει να συμφωνήσω σε αυτό. Και στο 12 ζητάει άρση ε, των, της εξαγοράς μέχρι να λυθούν όλες οι διαφορές. Κοιτάξτε, ε, ε, επειδή ο κάθε ένας εργαζόμενος μπορεί να υποβάλει κάποια αντίρρηση όσον αφορά την εξαγορά, δεν είναι δυνατόν να σταματήσει η διαδικασία. Δεν θα συμφωνήσω λοιπόν με τα 9, 10 και 12. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η εισηγήτρια θέλει να προσθέσει κάτι. Όχι. 9 Ιανουαρίου, προθεσμία υποβολής ε, των τροπολογιών 12 το μεσημέρι, επίσης στα αγγλικά οι τροπολογίες. 23-24 ε, ε, Ιανουαρίου θα μελετηθεί το ζήτημα και τον Φεβρουάριο θα έχουμε την συνέχιση. Πρώτο τελευταίο σημείο της μερισσίας διατάξεως κατάσταση διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο σχετικά με τους φακέλους με τους οποίους ε, συνεργαζόμαστε σε ενισχυμένη συνεργασία με άλλες επιτροπές. Ο κύριος Κόζα δεν είναι εδώ, επομένως το δικό του σημείο θα μας απασχολήσει άλλη φορά ε, και η κυρία Λαμπέρα δεν είναι εδώ. Ε, σχετικά με την ε, οδηγία για το ε, πρόγραμμα Δίκαιο και Ιθαγένεια 2012-2020. Δηλαδή είναι θέμα που μελετάει σήμερα η ΛΥΜΠΕ. Έχουμε όμως δύο εισηγητές που είναι εδώ και τους ευχαριστώ. Θα δώσω αμέσως το λόγο στην Λίζα Γιάκενσάρη για να μας πει που βρισκόμαστε όσον αφορά την πρόταση οδηγίας ε, σχετικά με τους ε, όρους ε, υποδοχής για τους για τις αποσπάσεις τις ενδομιλικές και υπαλλήλου, με υπαλλήλους τρίτων χωρών. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μάλιστα, όσον αφορά την οδηγία ECT, περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται για αποσπάσεις εσωτερικά μέσα σε ένα όμιλο η εταιρεία και πρόκειται για θέματα τα οποία είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών ΛΥΜΠΕ και της δικής μας ε, εδώ ομάδας. Και υπήρξαν αρκετές ε, διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ μας και καταλήξαμε, ε, καταφάνηκε το εξής. Είδαμε ότι στο τέλος τέλος, σε σχέση με τις δικές μας αρμοδιότητες, υφίσταται ένα μείζον πρόβλημα όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων. Πρέπει να καλυφθεί αυτό. Πρέπει να έχουν την ίδια αντιμετώπιση, την ίδια μεταχείριση οι εργαζόμενοι αυτοί, άσχετα από την προέλευσή τους. Ίδια αντιμετώπιση. Έχουμε ισχυρή εντολή. Και διαπίστωσα, αυτό ήμουν υποχρεωμένος να κάνω, το Συμβούλιο και εμείς ως Ευρωβουλή τις ίδιες ανησυχίες, ε, τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Θέλουμε η οδηγία να μην αποτελέσει αντικείμενο κατάχρησης. Γι' αυτό αναζητήσαμε ένα συμβιβασμό, σύμφωνα με τον οποίο όλοι οι εργαζόμενοι πραγματικά θα έχουν ίσα δικαιώματα. Θα απολάβουν ίσων δικαιωμάτων. Ένα δεύτερο σημείο για ε, ζωντανές έντονες συζητήσεις και για την αναζήτηση συμβιβασμού είναι ο καθορισμός ε, όσον αφορά ε, για παράδειγμα της διαχείρισης ε, και το Συμβούλιο θέλει να συνεχίσει δίνοντας συνέχεια στα πράγματα με βάση τα σημερινά πλαίσια ή τη σημερινή βάση με την υποβολή προτάσεων κτλ. Με τη βοήθεια για κολίνο εμείς προσπαθήσαμε να προσπίσουμε τη θέση του Κοινοβουλίου. Βρίσκονται υπό εξέλιξη αυτές οι διαπραγματεύσεις και συνεχίζονται. Και τα συμβαλόμενα μέρη γνωστοποίησαν ε, το ένα στο άλλο τις θέσεις τους. Ε, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει κανείς λόγο για πρόοδο ακόμα. Δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή λόγος για πρόοδο. Όμως, από την άλλη πλευρά, όπως και να έχει το πράγμα, οπωσδήποτε, εγώ σίγουρα θα με μεριμνήσω και θα δώσω αγώνα για τη δική μας θέση να είναι σεβαστή. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία λοιπόν. Καλή συνέχιση και καλό κουράγιο για τη συνέχεια που θα έχετε. Είναι θέμα το οποίο δεν μας απασχόλησε για πολύ καιρό, αλλά παραμένουν οι δυσκολίες και βασιζόμαστε πάνω σας και στην αποφασιστικότητά σας για να το προωθήσετε άλλη διαπραγμάτευση. Σέρτζο Κομφεράτη για την πρόταση οδηγία σχετικά με τις σε εισόδου και διαμονέ ε, εποχικών εργαζομένων προερχομένων από τρίτε χώρε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Ο τριμερή διάλογο ξεκίνησε χθε μόλι. Και πρέπει να πω στου συναδέλφου ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Δηλαδή, Έχουμε δυσκολίες στην επαφή μας με το Συμβούλιο, το οποίο θέλει να προτείνει λύσεις οι οποίες μπορούν να τροποποιήσουν εντελώς τον χαρακτήρα της οδηγίας από, εποχικό, από οδηγία εποχικής εργασίας να οδηγηθούμε σε οδηγία για ε, εργασία περιορισμένου χρόνου, χωρίς όρια και χωρίς περιορισμούς. Ε, θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Βεβαίως έχουμε εδώ σύμμαχο την ε, Κομισιόν. Η εργασία που έχει γίνει μέχρι τώρα υποβάλλει επιχειρήματα τα οποία ήταν περισσότερο ε, θέματα ΛΥΜΠΕ και η έκθεση Μωράης είναι εξαιρετική έκθεση που αποτελεί ε, σημαντικό βοήθημα στη συζήτηση. Μετά το πέρας των χθεσινών εργασιών νομίζω ότι δώσαμε στο Συμβούλιο και την Κομισιόν πολύ ενδιαφέρουσες ενδιαφέρουσες ε, για την κατεύθυνση την οποία θέλουμε να ακολουθήσουμε. Ε, μπούσουλας δικός μας βεβαίως είναι και ε, το κείμενο το οποίο είχαμε εγκρίνει στην Επιτροπή μας. Φυσικά θα πρέπει, αν θέλουμε να συνεχίσουμε με κάποιες πιθανότητες επιτυχίας, ε, θα πρέπει όλοι οι συνάδελφοι που ήταν σκιώδεις εισηγητήσεις στην προηγούμενη συζήτηση να έρθουν σε επαφή μαζί μας έτσι ώστε να ε, ε, βλέπουμε πώς προχωρεί η συζήτηση και ποια είναι τα σημεία διαμεσολάβησης τα οποία, επί των οποίων μπορούμε να συμφωνήσουμε. Η αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολη, αλλά νομίζω ότι η καλή σχέση μεταξύ των δύο επιτροπών βοήθησε τα σε αυτή την πρώτη φάση, έτσι ώστε να τεθεί σε σωστές βάσεις οι συζητήσεις και να μην αφαιθεί κανένα περιθώριο σε όσους, όπως η Επιτροπή, θέλει να τροποποιήσει την ουσία και την φύση της οδηγίας. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Χαιρετίζουμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα που μας είπατε. Ευχαριστούμε για τη σύνοψη που μας κάνατε και ευχαριστούμε βεβαίως ε, που υπεραμείνεστε των θέσεων της Επιτροπής μας. Με κάποια καθυστέρηση για την οποία ζητώ συγγνώμη από τους ε, ε, εμπειρογνώμονες φτάνουμε λέω στο σημείο 13 στη δημόσια κρεώαση που θα θέλαμε βάσει της Εκθεση ε, πρωτοβουλίας της Κέριμ Τελή όσον αφορά την κοινωνική στέγαση που αποτελεί δυνατότητα διεξόδου από την κρίση. Θα, μέσω, θα δώσω αμέσως το λόγο στην εισηγήτρια έτσι ώστε να κάνει την εισαγωγή την κυρία Καρυμαντελή και μετά θα δώσω το λόγο και στους ε, εκπροσώπους, ε, του, τους εμπειρογνώμονές μας αλλά και στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. κυρία Καρυμαντελή, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε αυτή την ε, ακρόαση και σας τους ειδικού που δεχτήκατε να έρθετε για να μας διαφωτίσετε με τις γνώσεις σας. Εγώ με τη διά μου δουλειά θέλω να δείξω πόσο η κοινωνική κατοικία μπορεί να αποτελέσει έναν μοχλό για να βγούμε από την κρίση. Η Ευρώπη ζει μια μεγάλη κρίση κατοικίας, η οποία μεγαλώνει. Και παρά τις αντιδράσεις της κοινή γνώμης, ιδιαίτερα το χειμώνα, που καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση για τους άστεγους είναι και απαράδεκτη, αλλά και πολύ δύσκολη. Η κατάσταση πήγε. Πήγε να επενδύσουμε στην κοινωνική κατοικία. Υπάρχουν κοινωνικές διαφορές, οι οποίες επιδεινώνονται. εκατομμύρια Μιλάμε μάλλον για 100.000 ε, άστεγους οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι στις απειλές που όλοι γνωρίζουμε στην Ευρώπη. Τα νίκια αυξάνονται. Η κατοικία τίθεται υπό δύσκολη κατάσταση δεν υπάρχουν αρκετά καταλήμματα για τους ανθρώπους αυτούς που δεν έχουν πολλά να πληρώσουν, οπότε το θέμα μιας αξιοπρεπούς κατοικίας είναι πολύ σημαντικό, γιατί όποιος δεν έχει στέγη, δεν έχει πρόσβαση ούτε σε ένα σωρό άλλα αγαθά. Και ειλικρινά θλίβομαι για την πολιτική ορισμένων χωρών που μειώνουν τελικά τις κοινωνικές κατοικίες και άρα πλήττουν έτσι και την συνοχή. Η κοινωνική κατοικία είναι κάτι το οποίο ζητάμε εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που να βασίζεται σε αρκετά μεγάλη προσφορά. Χρειαζόμαστε συνεπώς μέσα για να καταπολεμήσουμε ε, την ε, σπατάλη ενέργειας, να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που έχουν ορισμένοι να πληρώσουν για την ενέργεια και να ενισχύσουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για να αντιμετωπιστεί το θέμα της στέγης. Να επενδύσουμε στην κοινωνική κατοικία, αυτό σημαίνει ότι δίνουμε μια απάντηση και στο θέμα της γύρανσης του πληθυσμού και στην εξάρτηση των ηλικιωμένων ατόμων. Αλλά απαντάμε έτσι και στο δράμα που ζουν μερικές φορές οι νέοι, οι ομάδες που βρίσκονται στο περιθώριο και βέβαια οι άστεγοι. Επίγει είναι κοινωνικό το θέμα, αλλά όχι μόνο, είναι και οικονομικό βέβαια. Γιατί η κοινωνική κατοικία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο προκειμένου ε, να έχουμε μακροοικονομικά μια σταθερότητα. Αν υπάρχουν αρκετές κοινωνικές κατοικίες, τότε ε, μειώνεται ο κύκλος που οδηγεί τελικά σε ε, φούσκες στεγαστικές όπως το είδαμε στην Ισπανία. Η επένδυση στην κοινωνική κατοικία πρέπει να λαμβάνετε περισσότερο υπόψη στα διάφορα συστήματα επίβλεψης τα μακροοικονομικά. Έπειτα αποτελεί και μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης η επένδυση στη στέγαση. Είναι κάτι θετικό για την απασχόληση, είναι κάτι καλό για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, είναι καλό για τα νοικοκυριά, άρα είναι κάτι θετικό για τους Ευρωπαίους πολίτες. Μειώνεται έτσι ο ενεργειακός λογαριασμός που παίρνουν τα νοικοκυριά. Άρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα διορθωτικά ταμεία, δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να ενισχύσουμε τις επενδύσεις στον τομέα της κοινωνικής κατοικίας. Με τα χρήματα αυτά μπορούμε να αναπτύξουμε αυτά που χρειαζόμαστε σήμερα, δηλαδή την συνεχή κατάρτιση, την επαγγελματική κατάρτιση, στη, για πράσινες θέσεις απασχόλησης, προκειμένου να έχουμε απασχόληση στην Ευρώπη. Χρειάζονται επενδύσεις, επαρκείς επενδύσεις για το επόμενο δημοσιονομικό πολιτές πλαίσιο και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα να πάνε στην κοινωνική κατοικία. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο της έκθεσής μου που προτείνω στην Επιτροπή μας. Από εκεί και πέρα περιμένω και άλλα σχόλια και παρατηρήσεις για να προχωρήσουμε. Υπενθυμίζω αυτό που είπα στην αρχή, ότι η κοινωνική κατοικία μπορεί να αποτελέσει μοχλό για να αντιμετωπιστεί η κρίση στην οποία όλοι βρισκόμαστε. Πρόεδρος, για να καταλάβουμε καλά ποια είναι τα ερωτήματα και τι περιμένουμε από εσά για να βοηθήσετε την Επιτροπή μας. Δεν ξεχνάω ότι η έκθεση αυτή πρωτοβουλίας ε, εξετάζεται εδώ στην Επιτροπή μας τώρα που βρισκόμαστε στο τέλος των διαπραγματεύσεων για το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Να δούμε λοιπόν πώς θα συμπεριληφθεί η κοινωνική κατοικία στα διάφορα κεφαλαία του. Έπειτα, η ίδια η Επιτροπή πολλές φορές καταγγέλει διάφορα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Ωραία, από σας λοιπόν περιμένουμε συγκεκριμένες απαντήσεις για το τι πρέπει να προτείνουμε εμεί τώρα ώστε να καταλήξουμε σε κάτι θετικό. Το λέω αυτό βέβαια ξέροντας ότι εσείς έχετε ετοιμάσει τις παρουσιάσεις σας. Δεν τις αλλάξετε τώρα. Η Κλέρου πρώτα απ' όλα λοιπόν που είναι γενικό Γραμματέας του Open Liaison Committee for Social Housing. Είναι κοντά και η οποία μας βοηθάει σε πολλές υποθέσεις που εξετάζει η Επιτροπή μας. Δέκα λεπτά έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Εισηγήτρια. Ε, Βεβαίω ε, έχουμε προετοιμάσει εκ των προτέρων ε, την παρέμβασή μα, αλλά μια και μου δώσατε συγκεκριμένε οδηγίε από 30 θα σα παρουσιάσω 10 διαφάνειε. Η ΣΕΚΟΝΤΑΣ είναι η οργάνωση η οποία ασχολείται με 25 εκατομμύρια, 25 εκατομμύρια μονάδες κοινωνικής ε, στέγασης και ε, ε, επίσης ασχολείται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε, αυτά, σε αυτές τις, τους μοχλούς της ευρωπαϊκής ανάπτυξης. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να υπενθυμίσω ένα ιστορικό γεγονός. Δηλαδή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα έπαιξε ε, πρόδρομο ρόλο όσον αφορά την κοινωνική στέγαση. Το 2005 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άνοιξε ε, το δρόμο, ζητώντας από το Συμβούλιο και την Κομισιόν να ξεκινήσουν ε, να βλέπουν τις δυνατότητες που θα είχαν τα διαφορετικά ταμεία για να καλύψουν κάποιες ενεργειακές ανάγκες της κοινωνικής στέγασης Πάντα το Κοινοβούλιο ήταν πρόδρομος λοιπόν και ε, επομένως δεν είναι δυνατόν να, ε, από την άλλη πλευρά να πούμε ότι μπορεί η κοινωνική στέγαση να ειδωθεί χωρίς ε, την ευρωπαϊκή της διάσταση. Η στέγαση αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη έχει γίνει ένα κυρίαρχο μέλημα των ε, πολιτών. Ε, η τελευταία έρευνα, δημόσια έρευνα που έγινε από το Ίδρυμα του Δουβλίνου ε, το έδειξε μάλιστα γιατί από τα τέσσερα μεγάλα συμπεράσματα ένα από τα συμπεράσματα ήταν ότι η στέγαση και η, και η ποιότητα της στέγασης γενικότερα στην Ευρώπη βελτιώνεται αλλά η ασφάλεια της στέγασης δηλαδή η βεβαιότητα της στέγασης ε, ε, είναι ένα ποσοστό το οποίο διαρκώς μειώνεται. Δηλαδή όταν κάνουμε την ερώτηση ε, τους επόμενους 12 μήνες είστε βέβαιοι ότι θα έχετε δυνατότητα να παραμείνετε σε καλές συνθήκες στέγασης, η απάντηση είναι όχι δεν είμαι βέβαιος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από κοινωνική πλευρά ε, το διακύβευμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερο ουσιώδε. Νομίζω ότι αυτή η ανασφάλεια ε, τη στέγαση είναι για μα ένα από τα ζητήματα τα οποία ε, θέλουμε να απαντηθούν στην έκθεση αυτή. Επίσης, Υπάρχει βεβαίως και ε, ο αντίκτυπος της ε, κρίσης και η κοινωνική στέγαση μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να αποτελέσει μοχλό εξόδου από την ε, κρίση, αλλά η αγορά ε, στέγης δεν ε, τρελάθηκε ξαφνικά από τη μία στιγμή στην άλλη. Εδώ η κρίση οφείλεται και είναι απόρρια 20 ετών αδράνειας πολιτικής όσον αφορά την κοινωνική στέγαση. Νομίζω ότι η Ευρώπη, ε, και αυτό είναι εγγενές πρόβλημα στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, δεν ασχολήθηκε με την στέγαση σε τιμή προσιτή, βλέπε στην κοινωνική στέγαση. 20 ε, χρόνια λοιπόν πολιτικών που ευνοούσαν στην ουσία ε, μόνο τους ιδιοκτήτες που κατοικούσαν στο ιδιόκτητο ακίνητό τους. Επομένως, ακριβώς ε, μετά από 20 χρόνια ε, ε, κακών πολιτικών, το πρόβλημα βεβαίως έχει διονγκωθεί. Στις μελλοντικέ πολιτικές θα πρέπει να μην λησμονούμε ότι μια πολιτική στέγασης είναι μια πολιτική η οποία θα δώσει αποτελέσματα σταθερής και προσιτή στέγασης μετά από 20 βλέπε 30 χρόνια. Η καταπολέμηση της ένδυας βεβαίως είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μεγάλο μεγάλο διακύβευμα και αυτό, μεγάλη πρόκληση ε, της ε, κοινωνίας ε, και η πραγματογνωμοσύνη μας καταδεικνύει ότι εάν υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν έχουν ακόμα συζητηθεί αρκετά, είναι η καταπολέμηση της της ε, ενεργειακής αβεβαιότητας. Ε, δηλαδή, ε, εάν πέρα από το ενίκιο, πέρα από το κόστος στέγασης που πρέπει να καταβάλει κανείς, υπολογιστεί και αυτό το δεύτερο κατά κάποιο τρόπο ενίκιο, το οποίο αφορά την, την πληρωμή της ενέργειας, τότε πραγματικά... Ε, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η Κομισιόν μας λέει ότι θα δουλέψει ε, για τα θέματα αυτά για να ε, οδηγηθεί σε, μια ευρωπαϊ... σε έναν ευρωπαϊκό ορισμό του ευάλωτου καταναλωτή εντός εισαγωγικών, τον οποίον θα βοηθήσει με διάφορες πολιτικές. Δηλαδή μπορούμε να φανταστούμε ένα είδος ενεργειακής ασπίδας έτσι ώστε ε, όλοι οι καταναλωτές να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στην ενέργεια. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε εδώ και άλλους ορισμούς ε, για ε, ευάλωτους καταναλωτές, νέες κατηγορίες κτλ. Αλλά δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε και την κοινωνική κατάσταση. Η αγορά ενέργειας λοιπόν ε, που διέπεται και από ε, ευρωπαϊκές ε, οδηγίες, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και κάτι άλλο, για το οποίο ο πρόδρομος υπήρξε πάντα το Κοινοβούλιο και που άλλαξε την, τον ευρωπαϊκό τρόπο σκέψης. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν να αυξηθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα της στέγασης. Υπενθυμίζω ότι εάν θέλαμε να, αν, και αν μπορούσαμε να, να πάρουμε την απόφαση να ανανεώνουμε κάθε χρόνο 3% ε, του στόλου, κατά κάποιο τρόπο του στεγαστικού στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δημιουργούσαμε κάθε χρόνο 1,5 εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και μια νέα δυνατότητα πέραν των δυνατοτήτων που έχουν τα διορθωτικά ταμεία ε, και αυτό το συζητήσατε εσείς στα πλαίσια της συζήτησης για την ενεργειακή, ενεργειακή αποδοτικότητα. Ε, η δυνατότητα που δίνει ε, είναι μια δυνατότητα που δίνει το άρθρο 7, παράγραφος 7 και ε, που αφορά την δυνατότητα ε, μείωσης ε, του κόστους της ενέργειας σε συνεργασία με τα διευθυντικά ταμεία ή οποιαδήποτε άλλα υπάρχοντα εργαλεία κρατικής βοήθειας κτλ. Αναφέρεται σαφώς το, στο άρθρο 7, παράγραφος 7, αυτή η δυνατότητα καταπολέμησης της ενεργειακής ε, ε, αβεβαιότητας. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει ένα ε, συγκεκριμένο οικονομικό μοντέλο που να λειτουργεί και που να μπορεί η ενεργειακή το ενεργειακό κόστος, το κόστος της ενέργειας να αποζημιώνεται, να αποσβαίνεται από μόνο του. Όμως και δεν είναι δυνατόν να βασιστούμε σε ανθρώπους που δεν μπορούν να πληρώσουν για την ενέργεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, υπάρχει μία ιδιαίτερη χρηματοπιστωτική μόχλευση έτσι ώστε να βρεθούν χρήματα ε, για να καλυφθεί αυτό το κόστος το οποίο δεν μπορούν οι ίδιοι οι καταναλωτές να καλύψουν. Τέλος, γιατί δεν έχουμε και πάλι πολύ χρόνο, θα ήθελα να περάσω το κεντρικό μήνυμα, δηλαδή να φανταστούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε όντως να ε, επενδύσει άμεσα ή έμεσα έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη προσφορά προσιτής στέγης. Κάποιες ε, χώρες έχουν λάβει και συγκεκριμένες συστάσεις ε, από την αγορά στέγασης τους που και προβλήματα παρουσιάζει και μεγάλη αστάθεια η οποία οδηγεί και σε μεγάλη οικονομική αστάθεια. Οι συστάσεις ε, λοιπόν τις, ε, που περιέχονται στην πρόταση είναι πολύ στοχευμένες ε, σε πολλές περιπτώσεις αλλά δεν απαντούν τελικά στο μόνο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί τώρα. Δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε το κόστος ε, της στέγασης να γίνει προσετό, έτσι ώστε να υπάρχουν στην αγορά στέγης ε, ε, κατοικίες τις οποίες κανείς να μπορεί να καταλάβει με προσιτή τιμή. Έχουμε 110.000 110.000 ε, νέες ε, ε, στέγες, ενώ οι ανάγκες στέγασης αναφέρονται σε 390.000 νοικοκυριά. Επομένως, λείπουν περίπου 250.000 κατοικίες και αυτό στην έρευνά μας που έγινε μόνο στην, και αφορά μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως, νομίζω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να είναι πιο παρούσα ε, στις επενδύσεις για κοινωνική στέγαση και, εν πάση περιπτώσει, εάν πραγματικά θέλουμε να γίνει σταθερή η αγορά στέγης, ε, θα πρέπει να δεκαπλασιάσουμε την δυνατότητά μας να παράγουμε προσιτή στέγη. Ευχαριστώ πολύ και θα δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Μπάρμπαρα Στένμπεργεν, η οποία είναι η υπεύθυνη, επικεφαλής μάλλον, του Liaison Office της Διεθνούς Ένωσης των Ενοικιαστών. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που μας δώσετε την ευκαιρία να έρθουμε στην Επιτροπή σας. Εκπροσωπούμε 68 οργανώσεις από ολόκληρο τον κόσμο και εδώ θα μιλήσω εκ μέρου των καταναλωτών θα έρθω μετά σε κάποια μοντέλα για τους καταναλωτές, γιατί αυτό κάνουμε εμείς σε καθημερινή βάση. Δίνουμε νομική αρρωγή σε νοικιαστές, σε καταναλωτές και θέλω να πιστήσω λίγο την προσοχή σας σε αυτήν την πτυχή της αγοράς. Αρχίζουμε το δικαίωμα στη στέγαση. Πρέπει να αναγνωρίσουμε όλοι ότι η στέγαση είναι θεμελιώδες δικαιώμα. Υπάρχει και νομική βάση από αυτού. Μερικές φορές το ξεχνάμε. Υπάρχει όμως. Στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων το δικαίωμα σε αρρωγή για κοινωνική στέγαση. Ο Επίτροπος για Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης είπε κάποια στιγμή, ιδιαίτερα σε στιγμές οικονομικής κρίσης, η ανάγκη στέγασης που υπάρχει για την Ευρώπη πρέπει να προστατευτεί. Δηλαδή το δικαίωμα αυτό πρέπει να το εξασφαλίζουμε. Υπάρχει και ένα άλλο θεμελιώδες ε, δικαίωμα από την Ευρωπαϊκή Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, άρθρο 31. Η κοινωνική χάρτα, συγγνώμη, που τη λέει, λέει ότι ο καθένας έχει δικαίωμα άσκησης του δικαιώματός του σε στέγαση. Και το δικαίωμα αυτό πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα συντάγματα των χωρών ε, μελών. Οπότε, αν μη τι άλλο, τα κράτη-μέλη πρέπει να νιώθουν ότι δεσμεύονται από την υποχρέωση αυτή που αναφέρεται στην ε, Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν χώρες-μέλη που δεν έχουν καν επικυρώσει ακόμα το κείμενο αυτό. Άρα, αν θέλετε να διορθωθεί η κατάσταση, τότε πρέπει να στηρίξετε τις ομάδες εκείνων ενοικιαστών καταναλωτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης. Η προλαλήσασα ξεκάθαρα αναφέρθηκε στην ανάγκη να κοιτάξει κανείς περισσότερο από κοντά την κοινωνική στέγαση, γιατί είπε ότι αποτελεί στοιχείο για συνοχή στην Ευρώπη. Κατά μέσο όρο, 30% ένα νοικοκυριό δίνει για τη στέγαση. Πολλές φορές 40% στα πιο φτωχά νοικοκυριά. Εμείς λοιπόν ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να κοιτάξουμε και να δούμε γιατί η στέγαση κοστίζει τόσο πολύ και πώ μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο συνολικά τελικά καταλαβαίνετε όταν μιλάμε για 40% και μιλάμε για 78 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν καταλαβαίνετε γιατί. Ακριβώς γιατί είναι τόσο υψηλές οι τιμές της στέγασης. Πώς μπορούμε να βγούμε από αυτή την παγίδα. Θα σας μιλήσω για ένα μοντέλο Tenure neutrality. Είναι μια τεχνική έκφραση ουδετερότητα στην ενοικίαση. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει δίκαια πολιτική στέγασης. Που με τη σειρά της σημαίνει ένα απλό πράγμα. Σημαίνει ότι η διοκτησία, η ενοικίαση, ή μένοντας χαρακτηριστικά σε κάποιο χώρο πρέπει να στηρίζεται εξίσου χωρίς καμία διάκριση. Είτε είσαι νοικιαστής δηλαδή, είτε είσαι ιδιοκτήτης, είτε ζεις ε, συνεταιριστικά σε κάποια κατοικία, για το κράτος πρέπει να είσαι το ίδιο πράγμα. Πολλές χώρες μέλη και άλλες χώρες ολόκληρο τον κόσμο στηρίζουν την ιδιοκτησία και όχι τους ενοικιαστές. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε, αυτόν, σε αυτή την ε, σκληρή νομοθεσία που με τη σειρά της οδηγεί στην αγορά στέγασης στην οποία δεν έχουν πρόσβαση πάρα πολλοί άνθρωποι. Μιλάμε εδώ πέρα για ορισμένες ομάδες, για νέους, για μετανάστες, για φοιτητές. Πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τη δικιά τους κατάσταση απέναντι στη στέγαση. Γιατί για να μπορεί κάποιος να αποκτήσει σπίτι, να γίνει διοκτήτης δηλαδή, πρέπει να είναι φερέγγιος, αλλιώς δεν του δίνει βέβαια δάνειο τράπεζα που σημαίνει ότι κάπως πρέπει να βοηθηθεί στην αρχή, είτε με την ε, κοινωνική στέγαση, είτε βοηθώντας τον σε κάποια συνεταιριστική κατοικία, κάπως. Χρειάζεται μια ασφάλεια. Κανένας δεν γίνεται από την άλλη μεριά ενοικιαστής αν δεν ξέρει ότι θα προστατευτεί από καταχρήσεις. Πολύ ψηλά ενίκια, για παράδειγμα. Κοιτάξτε τι γίνεται στην κεντρική και στην ανατολική Ευρώπη. Εκεί δεν έχουμε σταθερό σύστημα για την προστασία των ενοικιαστών. Άρα πολλά μένουν να γίνουν και στις χώρες εκείνες όπου υπάρχει ένας νόμος για σωστό νίκη, αυτές οι χώρες να βοηθήσουν τις άλλες χώρες, οι οποίες δεν έχουν ακόμα τέτοιο σύστημα. Επανέρχομαι τώρα σε αυτή την ουδετερότητα ενοικίασης που σας έλεγα πριν. Η στεγαστική πολιτική πρέπει να έχει ως στόχο κατάλληλη στέγαση, χωρίς να έχοντας υπόψη ένα ειδικό προφίλ ενοικίασης. 100% ιδιοκτησίας σπάνια ισχύει σήμερα στα αστικά κέντρα, αν μη Πάντα χρειάζεται κάποια βοήθεια είτε κάποια βοήθεια στο νίκη που πληρώνει κανείς. Αυτό σίγουρα ισχύει στις πόλεις. Τι μπορούμε να κερδίσουμε λοιπόν από καλύτερες οικονομικές συνθήκες στέγασης. Από τη Γερμανία έχουμε κάποιο παράδειγμα. Μια έκθεση θα δημοσιευθεί την επόμενη εβδομάδα από τη μεγαλύτερη στεγαστική τράπεζα της Γερμανίας. Ένα ευρώ επένδυση στην ενέργεια οδηγεί σε 4 με 5 ευρώ απόδοση. Έτσι λέει. Κάτω χώρες τώρα. Από την στατιστική τους υπηρεσία. Ένα δισεκατομμύριο επένδυση ευρώ οδηγεί σε ανάπτυξη 40% ναι, και επιπλέον απασχόληση. Κερδίζει και το κράτος από τέτοια επένδυση. Μιλάμε για επένδυση σε στέγαση, έτσι. Στο κάτω-κάτω παίρνει και φόρο για τις κατοικίες αυτές. Τελικά όλοι έχουν να κερδίσουν ε, επενδύοντας στη στέγαση. Πρέπει συνεπώς να επενδύσουμε στην στέγαση γιατί έτσι βελτιώνουμε και τις συνθήκες ζωής, αλλά και την απόδοση. Ενισχύουμε και την οικονομία. Είναι προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας. Τι πρέπει να κάνουμε? Είναι ξεκάθαρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητες, άρα μπορεί να κάνει. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να έχει πιο προοδευτικούς κανόνες. Ήδη χρηματοδοτεί τις υποδομές. Γιατί να μην χρηματοδοτεί και στέγαση για όλους. Τώρα κάνουμε διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό. Έχουμε και τα κοινωνικά ταμεία. Δεν θα έπρεπε να δούμε πώς μπορούμε να συμπεριλάβουμε τέτοια μέτρα. Και έχουμε και το ERDF, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, που και αυτό μπορεί να βοηθήσει. Πάντως, το κύριο στοιχείο που θέλω να κρατήσετε είναι το εξή. Υπάρχουν εμπόδια. Κυρίες και κύριοι, ευρωβουλευτές, εσείς μπορείτε να μας βοηθήσετε. Έχουμε την περίπτωση, την Dutch case όπως λέγεται, την Ολλανδική περίπτωση που έχει να κάνει με την στέγαση και έχει να κάνει με τον ορισμό όσον αφορά την κοινωνική στέγαση. Ποιος δικαιούται δηλαδή η κοινωνική στέγαση. Είναι καταστροφή ο ορισμός αυτός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι η κοινωνική στέγαση προορίζεται μόνο για ομάδες που ε, είναι σε μειονεκτική κατάσταση κοινωνικά. Χωρίς ε, δηλαδή εισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή τα μεσαία στρώματα δεν έχουν πρόσβαση. Ο ορισμός αυτός είναι λάθος. Ο ορισμός αυτός που έχει στο μυαλό της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν και σε ζητάω, όχι λίγα πράγματα, μεγάλα πράγματα, να αλλάξει αυτός ο ορισμός. Τέλος. Κοιτάξτε λίγο στην, ε, την ενίσχυση του μη κερδοσκοπικού τομέα. Φυσικά και υπάρχουν πολλοί ιδιωτικοί επενδυτές, ιδιώτες επενδυτές, ο ιδιωτικός τομέας που επενδύει. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως για τον μη κερδοσκοπικό τομέα που επίσης μπορεί να επενδύσει. Δεν θα σας μιλήσω για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, δεν θα σας μιλήσω όμως για τις βέλτιστες πρακτικές. Βγαίνει με το καλύτερο σύστημα. Μη κερδοσκοπική στέγαση, δηλαδή Δανία, Βερολίνο, Γαλλία και συνεταιριστικές κατοικίες στην Τσεχία. Να λοιπόν μερικά πολύ καλά παραδείγματα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Για να ολοκληρώσουμε τις παρεμβάσεις των εμπειρογνωμόνων θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ζουλίς Οπτεμπέκ, της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Διεύθυνση Ευρώπη 2020, Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης της Ένδυας. Ε, good evening, Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεν έχω προετοιμάσει παρουσίαση θα ήθελα απλώς ε, να κάνω τρία σύντομα σχόλια. Και βεβαίως μετά θα απαντήσω σε όποια ερώτηση προκύψει. Όπως Αυτό σημαίνει ότι προτιμάτε να μιλήσετε μετά τις παρεμβάσεις των μελών. Ναι, ναι, θα το προτιμούσα. Νομίζω και εγώ ότι είναι το καλύτερο, λέει η Πρόεδρος. Φίλιπ Μπινιόν. Yes. Ε, Uh, Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την κυρία Καρίμα Ντελή γιατί ε, προετοίμασε μια εξαίρετη απογευματινή συνεδρία. Ακούσαμε σήμερα ομιλητές τους ε, οποίους είχα την δυνατότητα ε, να δω και να υποβάλω ερωτήματα σε εκείνη την απογευματινή συνεδρία που είχε οργανώσει η κυρία Ντελή πριν από δύο εβδομάδες και ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό να πω δύο λόγια παρόλα αυτά. Νομίζω ότι με τον, τρόπο, με τον ίδιο τρόπο ξεκίνησα ε, και την προηγούμενη φορά πριν από δύο εβδομάδες. Ε, το δικαίωμα στη στέγαση ε, δεν είναι δυνατόν να είναι καθολικό. Δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι έχουν όλοι δίκαιο στη, δικαίωμα στη στέγαση ενώ αρνούνται να πληρώσουν το ενίκιο. Αλλά αυτή νομίζω είναι η μόνη αρνητική σήμανση που θα κάνω. Ε, πριν από δύο εβδομάδες συζητήσαμε πολύ το θέμα της ενεργειακής ε, ε, αποδοτικότητας και της ενεργειακής ασφάλειας. Έγινε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση σχετικά με το πώς μπορούμε να μοιραστούμε βέλτιστες ε, πρακτικές και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, ευρωπαϊκούς ε, πόρους για να βελτιώσουμε την δυνατότητα προσιτής στέγασης σε συνδυασμό και με την ενεργειακή απόδοση. Και βεβαίως διαρκώς το ζήτημα της λεγόμενης ε, ιδιοκτησιακής ε, ουδετερότητας προέκυπτε. Πώς μπορεί να ε, δώσεις κίνητρα στους ενοικιαστές για να πάρουν μέτρα για μεγαλύτερη ενεργητική απόδοση. Οι εταιρείες ενέργειας, οι ηλεκτρισμού χρηματοδοτούν τα, ε, τις επενδύσεις τους και μετά μέσω μειώσεων των χρεώσεων ε, επιστρέφουν κατά κάποιο τρόπο την επένδυση αυτή στους ε, χρήστες. Αυτό όμως είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Νομίζω ότι θα είναι λίγο προβληματικό το να κρατήσουμε αυτό το ζήτημα μέσα στα πλαίσια των ευρωπαϊκών ενωσιακών αρμοδιοτήτων. Βεβαίω, όπως είπα και προηγουμένως, θα μπορούσαμε να το κάνουμε μέσω μοιράσματο, ας πούμε, και ε, βελτίστων πρακτικών και μέσω εμπλοκή και των τραπεζών. Νομίζω ότι ένα άλλο ζήτημα το οποίο προέκυψε ήταν η διαφορετική πολιτική στέγαση και ε, η σύνδεση με την χωροταξιακή πολιτική. Είχαμε μία φούσκα στις διάφορε χώρε μέλη, είχαμε μία φούσκα ε, στον οικοδομικό τομέα στην Ισπανία πριν από λίγο καιρό ε, όπου ε, δημιουργήθηκαν ε, μεγάλα, εκπονήθηκαν μεγάλα προγράμματα, το οποίο δεν ήταν όμως και στέγασης ή κοινωνική στέγαση, ήταν απλώς επενδύσεις. Στην στην... Στο Ηνωμένο Βασίλειο βλέπουμε τα τελευταία δέκα χρόνια να υπάρχει μια τάση να ρίχνουν οι δημοτικές αρχές σπίτια τα οποία όμως ε, είναι ακόμα σε καλή κατάσταση. Αυτά βλέπουμε λοιπόν σε πολλές χώρες ε, ε, πολιτικές οι οποίες τελικά οδηγούν σε αντίθετα αποτελέσματα. Πρέπει να γίνουν μελέτες έτσι ώστε να δούμε ποιες είναι οι πραγματικά βέλτιστες πρακτικές. Ελπίζω ότι η διαδικασία θα είναι επικοδομητική. Μπορεί να πάρει λίγο χρόνο, αλλά είμαι αισιόδοξο ότι τελικά θα, το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σέρκας και μετά η κυρία Κοστέλο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ τις εμπειρογνώμονες που ήρθαν ε, εδώ. Εγώ είμαι σκιώδης εισηγητής από πλευράς των σοσιαλιστών. Γι' αυτό και θα ήθελα τις παρουσιάσεις σας αν μπορείτε να μας τις στείλετε. Γιατί για την ομάδα μου, όπως βέβαια και για όλους τους συναδέλφους εδώ στην Επιτροπή μας αυτή, το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και επιπλέον θα αποκτάει όλο και μεγαλύτερη σημασία όσο περνάει ο καιρός και οι κοινωνικές επιπτώσεις ε, γίνονται περισσότερο αισθητέ λόγω της κρίσης. δυστυχώς μέσα από την κρίση βλέπουμε όλες τις αντιφάσεις και όλα τα προβλήματα της κοινωνίας μας. Γιατί δεν πρόκειται μόνο για αυτούς που δεν τους αναγνωρίζουμε τα, ανθρώπι, τα θεμελιώδη τους δικαιώματα. Εσείς πολύ καλά αναφερθήκατε στο φαινόμενο αυτό. Και όντως υπάρχουν καταστάσεις εντελώς παράλογες, όπως στη χώρα μου, όπου πάρα πολλοί άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους. Και βέβαια, ένα μέρος της κρίσης οφείλεται στο ότι επί 20 χρόνια δεν υπήρξε στην Ισπανία μια λογική πολιτική στέγασης. Τι κάνανε, δεν υπήρχαν λεφτά, δίνανε ένα δάνειο στους ανθρώπους για να πάρουν το σπίτι τους, οπότε τελικά μετανεβαίναν οι τιμές αφού πολλοί κόσμος είχε δάνεια για να αγοράζει σπίτια, δημιουργήθηκε έτσι αυτή η φούσκα και να τα αποτελέσματα. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι εμείς, παρόλο που είναι αργά τώρα που ξεκινάμε, έστω και τώρα να προχωρήσουμε και να βρούμε μια απάντηση. Πέρα από την ιδεολογία που μπορεί να έχει ο καθένας, όλοι να δεχτούμε ότι η αγορά είναι ατελής και ότι δεν μπορεί να προσφέρει ικανοποιητικά σε όλους αυτό που θέλουν. Άρα χρειάζεται να προβλεφθεί και κάποια προστασία. Ένα ζήτημα θέλω να θίξω, κυρία Πρόεδρε, και να ρωτήσω. Μερικές χώρες δεν θέλουν να αντιδράσουν ή η Ευρώπη δεν θέλει να τις ενοχλήσει για να αλλάξουν την πολιτική τους. Ε, λοιπόν, αυτό πρέπει να αλλάξει. Η Ευρώπη πρέπει να έχει έναν κοινό παρονομαστή. Στόχος μας πρέπει να είναι να βελτιώσουμε την κοινωνική προστασία και όχι να την κατεβάσουμε στα επίπεδα των χωρών εκείνων που περιφρονούν την κοινωνική προστασία ή την αγνοούν. Η κοινωνική δικαιοσύνη πρέπει να υπάρχει, είναι κοινωνικό αγαθό. Η έκθεσή μας, όπως είπατε και εσείς, ας ελπίσουμε ότι θα αποτελέσει ένα βήμα προς τα μπρος, ώστε να πιστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να σταματήσουν τα λόγια και να αρχίσουν τις πράξεις. Τέλος, κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα με την ε, Καρίνα Ντέλη θα δουλέψουμε πολύ καλά. Η κυρία Καρίνα Ντάλη Α ελπίσω ότι θα κάνει όλα όσα λέει, α αλλάξει λίγο τις προτεραιότητέ της. Να μιλήσει πρώτα για τους ανθρώπους και μετά για τον πλανήτη. Εκεί θα συμφωνήσω 100%, μαζί της. Επιτρέψτε μου που κάνω αυτό το αστιάκι. Μη βάζει πρώτα τον πλανήτη και μετά τους ανθρώπους. Πρόεδρος, Καστελό τώρα. Και μετά θέλετε και πάλι το λόγο, κύριε Νταλή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και την εισηγήτρια και ε, τις παρουσιάσεις, τις καλεσμένες μας για τις παρουσιάσεις τους. Είναι αλήθεια ότι οι επιπτώσεις της κρίσης έχει σαν αποτέλεσμα οι άνθρωποι να γίνονται πιο ευάλωτοι. Και πολλοί άνθρωποι νιώθουν να φοβούνται μήπως χάσουν τα σπίτια τους. Όντως πρέπει να το προσέξουμε αυτό όλος ιδιαίτερος. Έχω διάφορες ερωτήσεις. Ποιε από αυτέ είναι για τις καλεσμένε μας, κάποιε για την εισηγήτρια. Είμαι δημοτικό σύμβολο ε, έξω από το Δουβλίνο και έχω κι εγώ εμπειρίες, κακές εμπειρίες όμως, συνεργασίας ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στον τομέα αυτό. Γιατί κατέρευσαν στην αρχή της κρίσης και άφησαν πάρα πολύ κόσμο σε τραγικές καταστάσεις που δεν μπορούσαν πια να ελπίσουν σε μια κατοικία. Η ιδέα ήταν συνεργασία ιδιωτικού δημοσίου τομέα. Ναι, αλλά αν εμείς θέλουμε ανάκαμψη, πρέπει να μιλήσουμε για οικονομική ανακάμψη, πρέπει να μιλήσουμε και για την απασχόληση και για την εκπαίδευση και για την ε, στέγαση. Ένα σωρό πράγματα δηλαδή. Συνέπώ κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται συντονισμός. Δεν μπορείς να πεις ότι θα φτιάξω κοινωνικές κατοικίε και τελείω απλώ θα το κάνω. Όσον αφορά τώρα την ενεργειακή απόδοση. Συμφωνώ με τη δήλωση της Βαρκελόνης των Δημάρχων και νομίζω ότι πολλές πόλεις και το Δουβλίνο έχει συνυπογράψει. Είναι ένα χρήσιμο μέσο για να πετύχουμε την ενεργειακή αυτή απόδοση. Τώρα θέλω να ρωτήσω και πάλι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρω ότι στην Ιρλανδία... Πάω πολύ γρήγορα, λέει ο Μιλήτρια. Συγγνώμη. Το ξέρω, πάντα μου το λένε. Προσπαθούσα να είμαι σύντομη, γι' αυτό, Πρόεδρε. Έλεγα λοιπόν για την οικονομική, μάλλον γενικά για την αναγέννηση κατά κάποιο τρόπο και της στέγης χρειάστηκε οικονομική. Έλεγα λοιπόν για τη δήλωση της Βαρκελόνης που πιστεύω ότι είναι καλή και ευτυχώς έχουν υπογράψει πολλές πόλεις. Τώρα, για την ενοικιαζόμενη κατοικία. Σε πολλές χώρες υπάρχουν διαφορετικές προδιαγραφές. Θα ήταν χρήσιμο αν μπορούσαμε να έχουμε κάποιες κοινέ ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Πολλοί άνθρωποι ζουν κάτω από τραγικές συνθήκες, συνήθως οι πιο ευάλωτοι βέβαια. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν προδιαγραφές για τα ενοικιαζόμενα καταλήματα. Και στην χώρα μου υπάρχουν οργανώσεις οι οποίες συνεργάζονται πολύ καλά με τις τοπικές αρχές και βελτιώνουν τις συνθήκες στέγασης. Πρόεδρος, ρωτώ την Επιτροπή, στο Σώμα των Επιτρόπων, πώς χειρίζεστε αυτά τα θέματα, επίτροποι δηλαδή, πώς τα χειρίζονται. Γιατί, καλά, θα μας πείτε για την καταπολέμηση της ένδυας, στα πλαίσια της στρατηγικής 2020, προσέχετε αυτά τα θέματα κλπ. κλπ. Υπάρχει όμως και επίτροπος ανταγωνισμού που στέλνει επιστολές παντού και ε, αμφισβητεί τις επενδύσεις στην κοινωνική στέγαση. Οπότε να μας πει η Επιτροπή. Αλλά τώρα η Κάρη Μανταλή και μετά θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι γιατί οι συνάδελφοι κατανοούν ε, την συλλογική προβληματική ε, της στέγασης. Έχω όμως αρκετά ερωτήματα. Δεν συμφωνώ πολύ με τον κύριο Σέρκας ε, όταν λέει ότι πρώτα πρέπει να είναι καλά για τους ανθρώπους και μετά για τον πλανήτη. Πρέπει να είναι και τα δύο μαζί ταυτόχρονα κύριε Σέρκας. Δεν γίνεται Δηλαδή ταυτόχρονα αγωνιζόμαστε και κατά των κοινωνικών αδικιών και κατά των λαθεμένων επενδυτικών επιλογών. Κυρίως όσον αφορά τώρα τη χρηματοδότηση όταν μιλάμε για χρηματοοικονομική μόχλευση υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες ε, για γεωθερμική ανακαίνιση χρησιμοποιούν ας πούμε ευρωπαϊκούς πόρους. Αυτό είναι καλό. Έχετε κάποια προγράμματα τέτοια τα οποία έχουν δημιουργήσει θέσει εργασία σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο. Έχετε δηλαδή κάποια συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία για να δείξετε αυτή την επίπτωση. Δεύτερον, σαν οργανισμός. Είπαμε, ναι, ότι υπάρχουν οικοδομικές φούσκες, το ξέρουμε, αλλά ποια είναι τα εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σήμερα. Ε, στήριξη των ε, ενοικίων, ας πούμε, ή κάτι άλλο. Έχετε στοιχεία απάντησης πέρα βεβαίως από, την, ε, ε, από το να, ευνοηθεί, να υπάρξουν ευνοϊκοί όροι για την ε, οικοδόμηση νέας στέγης. Υπάρχουν και κάποια άλλα, κάποιοι άλλοι τρόποι για να ενθαρρύνετε την αγορά. Και δεύτερον, η πρόσβαση στην κοινωνική στέγαση μπορεί να διευκολυνθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Οπεντομπέκα, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι γεγονός ότι στην προσπάθειά μας να μειώσουμε και να καταπολεμήσουμε ε, την ε, ε, φτώχεια, βεβαίως η κοινωνική στέγαση είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ταυτοχρόνως όμως πρέπει να πω ότι έστω και αν υπάρχει ε, δικαίωμα στην ε, στέγη, η, αυτή, αυτό το δικαίωμα δεν μπορεί να αποτελέσει νομική βάση για νέα ε, δράση. Η Κομισιόν δεν έχει έτσι πολλούς τρόπους για να πείσει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορεί δηλαδή να αναλάβει νομική δράση σε αυτήν την διαδικασία η κρατική επιδότηση τώρα δεν νομίζω ότι αποτελεί πρόβλημα. Ε, ε, είναι, ε, είναι στις εξαιρέσεις. Το Ολλανδικό παράδειγμα είναι ακραίο παράδειγμα κοινωνικής στέγασης, το οποίο ξέφυγε λίγο από έλεγχο και είναι γεγονός ότι και στην Ολλανδία, παρότι είναι τόσο μικρότερη χώρα, υπάρχουν οι ίδιες μονάδες κοινωνικής στέγασης με την Γερμανία. Δεν νομίζω λοιπόν ότι το παράδειγμα της ε, ε, Ολλανδίας ε, είναι κλασικό παράδειγμα ευρωπαϊκό. Και το γαλλικό παράδειγμα, τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Δυστυχώς <coughs> δεν μπορώ να σας πω γιατί δεν έχω ιδιαίτερη γνώση από αυτού. Πάντως υπάρχει Υπάρχει εδώ και η αναφορά στην γαλλική περίπτωση και νομίζω ότι αν έχετε κάποια θέση σαν γενική διεύθυνση, αυτό θα μας, η θέση σας αυτή θα μας ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Ναι, ξέρω ότι έχουν υπάρξει εξαιρέσεις όσον αφορά τη δημιουργία κοινωνική στέγασης, αλλά κάθε φορά που υπάρχει εξαίρεση ε, υπάρχει και ένα όριο το οποίο μπορεί κανείς να ξεπεράσει. Και γι' αυτό λοιπόν οι συνάδελφοι από τη Γενική Διεύθυνση ΚΟΜ πρέπει να το μελετήσουν το θέμα. Δεύτερον, δεύτερον η δεύτερη ιδέα, τα διαρθρωτικά ταμεία όλα αυτά ε, τα ταμεία δίνουν πολλές ε, δυνατότητες ε, για αύξηση του αποθέματος κοινωνικής στέγασης και για μείωση των λογαριασμών της ενέργειας. Υπάρχουν πολλά εργαλεία τα οποία είναι διαθέσιμα και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες μπορούν πολλά να κάνουν, αλλά βεβαίως για το ERDF και για το ESF ε, η συνολική χρηματοδότηση θα είναι γνωστή μετά το πέρας των χρηματοδοτικών ε, διαπραγματεύσεων. Εμείς έχουμε κάνει πρόταση, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας επίσης και μια άλλη, σε μια άλλη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία νέου ταμείου για την ευρωπαϊκή βοήθεια προς τους ε, ε, λιγότερο ευνοημένους. Ε, θέλουμε δηλαδή να βοηθήσουμε τους αστέγους να ξαναμπούν σε μια διαδικασία κανονικής στέγης κτλ. Εάν αυτό το πρόγραμμα και αν αυτή η πρόταση ε, γίνει δεκτή, τότε θα αλλάξουν πολλά όσον αφορά τα προβλήματα τα οποία συζητούμε τώρα. Επίσης, από όσο ξέρω, όσον αφορά την ίδια την κοινωνική στέγαση, δεν υπάρχουν ε, συγκεκριμένες ε, πρωτοβουλίες, δεν μπορώ να πω ενωσιακές, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Αυτά είναι τα σχολιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Μπορώ να σας πω, χωρίς πρώτερη διαβούλευση, ότι η ιδέα νέου ταμείου ε, για τους ε, ε, πιο φτωχούς που θα μπορούσε να βοηθήσει το πρόβλημα της κοινωνικής στέγασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ξέρετε πόσο πόσο κάτω είμαστε από το κατόφλι. Να συνεχίσω στα γαλλικά γιατί στα αγγλικά δεν μου βγαίνει, λέει η Πρόεδρος με τον προϋπολογισμό που έχετε προβλέψει ε, για θέματα κοινωνικής στέγασης ε, δεν ε, μπορούν να στηριχτούν ούτε καν σε λειτουργία τα κοινωνικά παντοπολία. Επομένως, με μεγάλη δυσπιστία βλέπουμε αυτά που λέτε. Αλλά βεβαίως σημειώνω την καλή βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ασχοληθεί με αυτά τα κοινωνικά ζητήματα. Αλλά πρέπει να είστε πιο συνεκτικοί και πρέπει να βρεθούν και άλλα χρήματα και άλλοι τρόποι. Θα δώσω τον λόγο για πέντε λεπτά ακόμα στην κάθε μία, στις δύο μιλήτρες. Ξέρω ότι είναι πολύ αγχωτικό αυτό, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα απαντήσω. Βέβαια, φαντάζομαι δεν υπάρχει δυνατότητα να επιστρέψουμε στις διαφάνειες μου. Όσον αφορά τις επιπτώσεις, να γίνουν δηλαδή περισσότερα πράγματα στο κοινωνικό επίπεδο και τη στέγαση. Μα ακριβώ αυτό βάζει και στο τραπέζι νέα πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Είναι διαφάνεια που θέλω να σας δείξω που λέει ότι σε πολλές μελέτες για τι επιπτώσει των προγραμμάτων όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση. Υπάρχουν προγράμματα σε διαφορετικές χώρες. Στην Τσεχία, όπου έγινε ένα πρόγραμμα για ηλιακού ηλιακούς στα ψηλακτήρια. Αν δείτε το πρόγραμμα αυτό, τι σκέφτεται κανείς. Δημιουργούμε θέσεις απασχόλησης για αυτούς οι οποίοι θα εγκαταστήσουν τα φωτοβολταϊκά στις σκεπές των κτηρίων. Όμως, η απασχόληση που δημιουργείται και καταστρέφεται στον ενεργειακό τομέα υπάρχει, αλλά το πιο σημαντικό είναι στις υπηρεσίες που είναι γύρω από το θέμα των φωτοβολταϊκών, γιατί πρέπει να γίνει και πολύ κοινωνική δουλειά και πριν και μετά για τη συντήρηση Άρα η ιδέα αυτή του προγράμματος ενεργειακής απόδοσης δεν έχει να κάνει μόνο με τα τεχνικά επαγγέλματα, έχει να κάνει γενικότερα με την απασχόληση γύρω από το θέμα. Όσο για τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ενοικίασης. Η στέγαση ε, βλέπετε είναι ένας τομέας στο οποίο το κόστος έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Διότι χρησιμοποιούνται νέα υλικά υψηλών προδιαγραφών που είναι ακριβά. Κάποιοι ανελκυστήρες για παράδειγμα ε, κατασκευάζονται σήμερα μόνο από δύο-τρεις εταιρείε γιατί μόνο αυτές ανταποκρίνονται στις πρόσφατες προδιαγραφές. Έπειτα. Του ποια μπορεί να είναι τα άλλα μέσα, γιατί δεν λειτουργεί η αγορά στέγασης, δεν προσφέρει. Και μας μας ενδιαφέρει προστασία των καταναλωτών. Σε χώρες όπως η Ισπανία και η Ουγγαρία, εκεί η... το σύστημα υποθήκευσης των σπιτιών έχει παγιδεύσει τους ανθρώπους συχνά για όλη τους τη ζωή. Και αυτό πρέπει να το δούμε, γιατί αν δεν έχετε επαρκή προστασία των καταναλωτών στην αγορά υποθηκών, τότε πλήττεται ο καταναλωτής. Υπάρχουν πάρα πολλές τράπεζες σε διάφορες χώρες που ο ισολογισμός τους δείχνει ότι έχουν πάρα πολλά περιουσιακά στοιχεία από τη στέγαση. Εκεί χρειάζεται κάπως καλή βούληση για να αλλάξουν τα πράγματα. Οι τράπεζες να μπορέσουν να μεταφέρουν τα ποσά αυτά, αλλά και χρειάζεται βέβαια διαπραγμάτευση μεταξύ τραπεζών και άλλα. Υπάρχει τρόπος όμως. Επίσης μπορούμε να βοηθήσουμε συνεταιρισμούς, ε, από κοινού ιδιοκτησίες που μπορεί να είναι εν μέρη κοινωνικές, εν μέρη όχι. Υπάρχουν πολλές λύσεις δηλαδή. Τέλος. Το θέμα της πρόληψης και καλύτερης δαπάνης ή τέλος πάντων πώς θα αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιτάει την αγορά τη στεγαστική ώστε να μην υπονομεύει τη δυνατότητα των καταναλωτών ε, να έχουν πρόσβαση σε ιδιόκτητη κατοικία. Στην έκθεση που θα ψηφίσετε, οι τροπολογία στην έκθεση Φερέρα, το θέμα είναι πώς θα αλλάξετε την λογική. Αν δείτε μόνο τις δαπάνες χρόνο το χρόνο, δεν θα οδηγηθείτε πουθενά. Στη στέγαση χρειάζονται επενδύσεις, επενδύσεις που αποδίδουν αργότερα. Το θέμα είναι πώς θα, γίνει, πώς θα γίνουν καλύτερες δαπάνες. Γιατί έτσι θα έχετε δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης στο μέλλον. Πολλές επικρίσεις ακούγονται για το γεγονός ότι η πρόσβαση στην κοινωνική κατοικία ε, δεν γίνεται πάντα με διάφανο τρόπο. Εντάξει. Υπάρχουν όμως νόμοι και υπάρχουν διαδικασίες. Τώρα, κατά πώς εφαρμόζονται, μερικές φορές πρέπει να διαλέξει κανείς ανάμεσα σε μία γυναίκα με τέσσερα παιδιά και μία γυναίκα με πέντε παιδιά. Αυτή είναι η επιλογή για την κοινωνική κατοικία. Ε, τι θέλετε να γίνει. Δεν έχω λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολλές ήταν οι ενδιαφέρουσες ε, συζητήσεις. Και αυτό δείχνει και πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Ε, ως εκπρόσωπος ενοικιαστών και καταναλωτών, εγώ θέλω, θα ήθελα διαφάνεια στην αγορά, γιατί θεωρώ ότι η διαφάνεια γιατρεύει τα πάντα, είναι πολύ καλό πράγμα. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε λίγο πώς χώρες ε, όπως ε, η Ελβετία ή η Αυστρία ή η Γερμανία με μεγάλο ποσοστό ε, προσφερωμένων προς ενοικίαση κατοικιών έχουν λύσει πολλά προβλήματα μέσω των, της ε, απόλυτης διαφάνειας. Μπορεί να δείτε ας πούμε στο στο διαδίκτυο να βρείτε ένα συγκεκριμένο σπίτι που είναι σε συγκεκριμένη πολυκατοικία, σε ένα συγκεκριμένο δρόμο του ωραίου Βερολίνου και να ξέρετε λοιπόν ακριβώς πόσο είναι το ενίκιο αυτό. Νομίζω ότι αυτό ε, έχουμε, έχουμε πληροφορίες και έχουμε δυνατότητα μάλλον να σας δώσουμε πληροφορίες σχετικά με το πόσο μπορεί ε, να εφαρμοστεί ένα σύστημα το οποίο το λέμε Μίτσπιγερ στα γερμανικά και το οποίο ε, ακριβώς δίνει τη δυνατότητα υπολογισμών ενοικίων επίσης ε, χρειαζόμαστε διαφάνεια για να δούμε κατά πόσον έχει επιστραφεί η επένδυση για ενεργειακή απόδοση. Εάν εξυγχρονιστεί ε, ένα κτίριο, μπορεί τότε η τιμή να είναι ε, ψηλότερη από ένα ε, άλλο κτίριο το οποίο δεν έχει εξυγχρονιστεί. Γιατί το κόστος της ενέργειας θα είναι πολύ μικρότερο και επομένως έχουμε ισορροπία τελικά. Και είναι αυτό το σύστημα της εξουδετέρωσης ας πούμε της διαφοράς του ενοικίου. Έχουμε ψηλότερο ενίκιο, το οποίο όμως, το οποίο όμως έχει ενσωματώσει το κέρδος του εξυγχρονισμού και της ε, ε, ενεργειακής, ε, βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης. Το ξαναλέω λοιπόν, έχουμε χαμηλότερο ενίκιο, αλλά αυτό έχουμε ψηλότερο ενίκιο και ενσωματώνεται εκεί και το κέρδος. Υπάρχουν ε, energy labels ε, στην Ευρώπη, έχουν ετικέτες ε, για την ενέργεια ενεργειακή απόδοση. Μην το λησμονούμε αυτό. Μπορούμε να τους σπρώξουμε λίγο έτσι ώστε να τους βρίσκουμε και πιο πολύ μπροστά μας στην αγορά. Αυτά ζητώ εγώ όσον αφορά την διαφάνεια λέτε έχουμε προβλήματα με τις ε, εταιρικές σχέσεις ε, δημοσίου και ιδιωτικού ε, τομέα. Εντάξει, υπάρχουν όμως εμπειρίες καλές σε πολλές χώρες. Νομίζω ότι οι εταιρικές σχέσεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα είναι ενδιαφέρουσες εάν έχουμε, αν υπάρχει ε, μάλλον εάν πρέπει να δημιουργηθεί εκ νέου ο τομέας κοινωνικής στέγασης. Ε, όμως ε, δεν αποτελούν αυτές οι συμπράξεις την ενδεδειγμένη λύση έτσι ώστε να βρεθούν λύσεις όσον αφορά μεγάλες ελλείψεις στέγης. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε και λίγο ε, το γιατί χρειαζόμαστε έναν, ένα τομέα στέγασης που δεν θα έχει ε, σαν κύριο και μοναδικό στόχο την, ε, το κέρδος. Το ίδιο γίνεται και με τα σχολεία. Το ίδιο, δεν ακολουθήσουμε λίγο το πρότυπο που ακολουθούμε με τα σχολεία, με τους ερφονιπιακούς σταθμούς, τα νηπιαγωγεία κτλ. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι ε, μη κερδοφο... μάλλον όχι, ε, ε, επενδύσεων οι οποίες δεν αποζητούν το κέρδος και που μπορούν να μπορεί να ακολουθήσει σαν πρότυπο, ας πούμε, η κοινωνική στέγαση. Στο Άμστερνταμ, στην Ολλανδία, ε, εάν θέλει κανεί κοινωνική στέγη θα πρέπει να περιμένει 12 χρόνια. μάλιστα. Τι κάνουν λοιπόν οι Ολλανδοί. Όταν τα παιδιά γίνουν 18 ε, ε, χρονών, τους κάνουν αμέσως, τους δηλώνουν έτσι για αυτήν την κοινωνική στέγαση, έτσι ώστε όταν πραγματικά χρειαστούν δικό τους σπίτι να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην κοινωνική στέγη. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει η Σα Ευχαριστούμε πρώτον τους διερμηνείς που μας ακολούθησαν μέχρι το τέλος αλλά βεβαίως και τις καλεσμένες μας, τις εμπειρογνώμονες, οι οποίες μας είπαν εξαιρετικά ενδιαφέροντα και σημαντικά πράγματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε ε, στην έκθεση πρωτοβουλία ε, που θα είναι πολύ σημαντική για την Επιτροπή Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων, να ξεκινήσουμε επιορθών βάσεων. Ποια άλλη επιτροπή μπορούσε να ασχοληθεί με το θέμα αυτό ε, και τελικά λέω ότι εμείς εδώ, εδώ στην Επιτροπή Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. 20 και 21 Φεβρουαρίου θα υποβληθεί η έκθεση. Θα είναι σύντομη η προθεσμία υποβολής τροπολογιών μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου. 20-21 Μαρτίου θα τις ε, μελετήσουμε. 22 Απριλίου θα μελετήσουμε τις, ε, τροπ, πόλο, ε, συγγνώμη, τις συμβαστικές τροπολογίες ε, και μετά θα περάσει την Ολομέλεια. Πολύ ωραία. Ε, λοιπόν, σας εύχομαι να περάσετε καλά ε, τις γιορτές και να γυρίσετε με χαρά στη δουλειά σας στις 14 Ιανουαρίου, οπότε και θα έχουμε στις 7 το απόγευμα της ιδίας αυτής μέρας στο Στρασβούργο έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ πολύ.